Ja, liebe Kolleginnen und... Αγαπητοί, αγαπητές και ένας αγαπητός υπάρχει, όχι, συνάδελφοι. Ξεκινούμε και πάλι τονίζω το αγαπητές συνάδελφοι, Τόμς, Κάπλ, Μπερές τώρα που έρχεται. Τέσσερις εκ των κυριών συναδέλφων μας βρήκαν το δρόμο μπορεί να εμφανιστούν και άντρες σύντομα στην Επιτροπή μας. Ερωτώ πάντως εάν έχετε αντιρρήσεις. Για την ημερήσια διάταξη όχι. Εγκρίνεται σημείο 2 στην ημερήσια διάταξη ανακοινώσεις. Θα ήθελα να σας ε, ενημερώσω για την αποφάση των συντονιστών, για τις αποφάσεις των συντονιστών 11 Ιουλίου. Καταρχάς, προτεραιότητα. Σε ποιους φακέλους θα, ε, θα δοθεί η προτεραιότητα με βάση τις προτάσεις των συντονιστών εκρίθη σκόπιμο να μην ληφθούν αποφάσεις ε, που θα χορηγούν προτεραιότητα σε κάποια θέματα και αυτό ισχύει για όλα πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, συνεργασία μεταξύ επιτροπών ε, στα, στα προγράμματα ανατομής και αποφασίστηκε να μην δοθεί γνωμοδότηση. Ωστόσο, θέλουμε η Επιτροπή μας να συμμετάσχει στην συνολική διαδικασία για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, πρόταση ψηφίσματος και τα θέματα τα σχετικά με τους τομείς μας. Για τους ορισμούς στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουμε σημειώσει τις θέσεις Πρόεδρου Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμφωνίου. Σχέδιο ε, συνεδριάσεων από τον Ιανουάριο στον Απρίλιο του 2019. Έχει εγκριθεί, το έχετε λάβει. Επίσης, συντονιστέ ασχολήθηκαν και με τις ε, αντιπροσωπείες για το δεύτερο έμισο του 2018. Αντιπροσωπεία με αποστολή στις Ηνωμένες Πολιτείες καταρχάς. Ε, συζητήθηκαν διάφορες τοποθεσίες και, διάφορα, και σχέδια προγράμματος χωρίς σχέδια, χωρίς σχόλια, συγγνώμη και αποφασίστηκε να μην επαναδιατεθεί η θέση που είχε προβλεφθεί για την ομάδα ECR. Κίνα, προσχέδιο προγράμματος, προτάσεις θα κατατεθούν έως την εβδομάδα υπαριθμών 29 το αργότερο. Το ίδιο και για την αντιπροσωπεία στην Ιταλία. Οικονομική διακυβέρνηση επίσης. με τους διοικητικού διευθυντή και αναπληρωματικό ε, διοικητικό διευθυντή συμφωνήσαν οι συντονιστές πώς θα προχωρήσουν επίσης ε, συνάντηση με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων 8-9 Οκτωβρίου για την Ελλάδα θα μπει το θέμα στις ε, ημερήσιες διατάξεις και στους συντονιστές αλλά και στην FAWG, στην ομάδα εργασίας δηλαδή. Στη συνέχεια αποφασίστηκε να μην γίνει η συνάντηση εποπτείας της, στην ε, συνεδρία 8 Οκτωβρίου, αναφορές καλούνται οι συντονιστές να στείλουν σχόλια ε, το αργότερο στην εβδομάδα με αριθμό 29. Συντονιστές, ε, λοιπά θέματα, συγγνώμη, διάφορα. Οι συντονιστές συμφωνούν να συμπεριλάβουν στην προσεχή μερική διάταξη το, το σημείο 1697 του 2016 συμπεράσματα, τελικά συμπεράσματα της έρευνας του διαμεσολαβητή αυτά για τις ανακοινώσεις του Προέδρου και μπορούμε να ξεκινήσουμε στην ημερήσια διάταξη το σημείο 3 σχέδιο γνωμοδότησης για, την, ε, για τις συνέπειες ορισμένων πλαστικών στο περιβάλλον έχουμε εδώ υποχρέωση μόνο για γνωμοδότηση η ένβη είναι κατ' ουσίαν αρμόδια σε ενημερώνω δε ότι πρέπει 24 ε, Σεπτεμβρίου δεδομένων των στενών χρονοδιαγραμμάτων της ε, κατουσίαν αρμόδιας ΕΝΒΗ να ψηφίσουμε τη γραμμοδότηση αυτή και τώρα έχουμε αυτή τη γραμμοδότηση με την κυρία Μπάρβαρα Κάβολ, συντάκτρια. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ο περιορισμός των ε, συνεπειών των των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον ε, είναι το θέμα της έκθεσής μας. Αφορά κυρίως τα πλαστικά τα οποία ε, απειλούν τα οικοσυστήματα, τα θαλάσσια, την δημόσια υγεία, τον τουρισμό, την αλία, την αυσιπλοεία με προβλήματα τα οποία γνωρίζουν ε, όλοι με 18 κύριους ε, ρηπαντές όπως ε, την Κίνα, τις Φιλιππίνες, το Χονγκ Κόνγκ αλλά και τις Ηνωμένε Πολιτείε, και 80% των ε, θαλάσσιων πλαστικών αποβλήτων προέρχονται από αυτά τα 18 κράτη. Με πρώτο συμπέρασμα λοιπόν δικό μου την προσπάθεια για την αποφυγή της θαλάσσιας ρήπανσης για την οποία χρειαζόμαστε την συνεργασία των πάντων και της ε, ομάδας των 7, των 8, των 20 ε, των διεθνών οργανισμών. Πρώτη παρατήρηση αυτή λοιπόν και δεύτερη χρειάζεται να ενισχυθεί η κυκλική και η οικονομία της ανακύκλωσης με ποσοστά μόνο 10% οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα καθώς μένουν μεταξύ των κύριων ε, υπέτειων για τη θαλάσσια ρήπανση. Πρέπει λοιπόν να μειώσουμε και να απαγορεύσουμε σε σημαντικά ποσοστά την παραγωγή και απόρριψη πλαστικών στις θάλασσες. Έχουμε μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στηρίζεται σε μια έρευνα που καταγράφει και τα πλαστικά μίας χρήσης ε, που κατά κύριο λόγο είναι μπέτια για τη ρήπανση, όπως γόπες τσιγάρων και ε, διάφορα άλλα μικρό αντικείμενα, τα οποία αποτελούν συνολικά το, οι σακούλες ε, πλαστικές κτλ, τα οποία παρτίζουν τα το 70% των θαλάσσιων ε, απορριμμάτων. Πρέπει να μειωθεί λοιπόν ε, η απόρριψη τους κατά 50%. Πρέπει να υπάρξει μια απαγόρευση της παραγωγής τους ώστε να ενισχυθεί ο περιορισμός ε, της χρήσης και να αναλευθούν μέτρα σχεδιασμού που να, που να επιτρέπουν την αποφυγή της χρήσης αυτών των ε, πλαστικών μιας χρήσης, όπως σε παραδείγματι είναι τα καλαμάκια στα πλαστικά ποτήρια. Θα έχουμε την κάλυψη του κόστους σε μεγάλο ποσοστό από τις ε, εταιρείες που παράγουν. Θα έχουμε ένα σημαντικό ποσοστό εξοικονόμησης για την παραγωγή, για τον καταναλωτή και για την ε, αλληλεία, καθώς θα αυξηθούν τα έσοδά της. Υπάρχει ωστόσο μία ένα σημείο το οποίο έχει να κάνει με τη μετακύληση του κόστου στον καταναλωτή και σε αυτό θέλω να σταθώ με την τρίτη μου παρατήρηση γιατί πρέπει να κοιτάξουμε την αναλογικότητα ε, στην χρήση. Το 50% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ε, αυτά τα πλαστικά είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Υπάρχει ανάγκη να βρεθεί για την διευκόλυνση τους μια νέα λύση ε, και η ε, δυνατότητες που προβλέπονται για την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν για τις επιχείρησεις αυτές δεν είναι ικανοποιητική. Χρειάζεται λοιπόν μια αξιολόγηση συνεπειών ώστε να υλοποιηθεί ουσιαστικά η αναλογικότητα. Πιο αυστήρες προδιαγραφές ε, και ε, ξεκάθαρα στοιχεία για, τις, για τα προϊόντα που είναι βιολογι, βιο, αποδομήσιμα στη θάλασσα, αλλά και νέες στρατηγικές που θα επιτρέψουν μέσα στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να καλυφθούν οι ανάγκες και σε οικονομικούς όρους ώστε να μην πληγεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Εάν λοιπόν μπορέσουμε να τη στηρίξουμε θα έχουμε όχι μόνο ε, αποφύγει την απώλεια ανταγωνιστικότητας αλλά και δημιουργήσει 30.000 θέσεις εργασίας επιπλέον. Ένα άλλο ζήτημα, μια μια άλλη διαπίστωση για μένα είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο την ευαισθητοποίηση και την συμμετοχή του ίδιου του πολίτη στην διαχείριση των αποβλήτων, στην ε, ανακύκλωση, στην διαλεκτική απόρριψη και νομίζω ότι αυτό ε, είναι ένας στόχος που μπορούμε να επιδιώξουμε περισσότερο. Με πολύ μεγάλη χαρά συνεργάζομαι με τους χειώδεις ηγητές για να συγκεκριμενοποιήσουμε τις ε, τροπολογίες και περιμένω τις επόμενες συνεδριάσεις μας ώστε να δώσω πιο συγκεκριμένε προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ την εισηγητρία. Κυρία Τόμς Ελκ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κάπελ για το έργο της. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο αποτελεί μεγάλη πρόκληση ε, για τον κλάδο. Πράγματι έχουμε και νέες προκλήσεις αλλά και νέες ευκαιρίες η Ευρώπη μπορεί και πάλι να βρεθεί σε ηγετική θέση και στον, ε, από πλευρά κλάδου. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα, αλλά ακόμα περισσότερο να δράσουμε. Η οδηγία για τα πλαστικά είναι μια καλή πρόταση για το περιβάλλον και για το μέλλον μας. Όμως, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτός ε, ο τομέας της ε, διάθεσης πλαστικού στο περιβάλλον είναι ένας ε, τομέας περίπλοκος και απαιτεί μια ε, πολύπλευρη προσέγγιση από όλες τις ομάδες και από τον κλάδο και από τους καταναλωτές. Η ομάδα μου είναι στηρίζει την απαγόρευση των πλαστικών μίας χρήσης, αλλά χρειαζόμαστε ένα περιθώριο, ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής, ιδίως ό,τι αφορά τις συσκευασίες. Επομένως, χρειαζόμαστε ε, συσκευασίες που θα είναι οικονομικά αποδοτικές, δεν θα έχουν δηλαδή και πολύ μεγάλο κόστος και για τον ίδιο τον καταναλωτή και το καθεξής. Εάν ο κλάδος δεν είναι ακόμα σε θέση να μας δώσει την ποιότητα που χρειαζόμαστε, πρέπει να δώσουμε το απαραίτητο χρονικό περιθώριο. Αλλά είμαι βέβαιη ότι αυτό ε, θα μας βοηθήσει να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Όμως και πάλι χρειάζεται και ο κλάδος ένα χρονικό περιθώριο για να προσαρμοστεί. Τώρα, να σταθώ στο ζήτημα της ε, παιδεία και της ε, ενημέρωσης ε, των καταναλωτών. Είπε η κυρία Κάπελ ότι τα περισσότερα απορρίμματα δημιουργούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρεθεί σε αυτή την ε, προεξάρχουσα θέση και εντός αλλά και εκτός. Να στείλουμε αυτό το μήνυμα ότι όλοι ανά τον κόσμο θα πρέπει να φροντίζουν το περιβάλλον, ότι έχουμε μόνο έναν πλανήτη και θα πρέπει να τον φροντίζουμε. Τέλος, θα πω ότι είμαστε υπέρ της απαγόρευσης ε, των πλαστικών μίας χρήσης, αλλά χρειάζεται μια πολύπλευρη προσέγγιση και θα πρέπει να δώσουμε το το χρονικό περιθώριο προσαρμογή ε, στον κλάδο. Ευχαριστώ. Ähm, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τόμς. Κύριος Λούκε, ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Κάπελ, τη συντάκτρια, για την ε, Πολύ σημαντική αυτή η έκθεση που μας παρουσίασε σήμερα. Συμμερίζομαι τα σχόλιά της. Έχω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις να κάνω για να εμπλουτίνουμε την ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής μας. Έχουμε εδώ να κάνουμε με έναν προβληματισμό που έχει και οικονομικά χαρακτηριστικά, όχι μόνο περιβαλλοντικά και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει τη δυνατότητα η Επιτροπή μας να διατυπώσει τις θέσεις της προτείνοντας κατάλληλες λύσεις για το πρόβλημα της ρήπασης της θάλασσας και της απορρίψης πλαστικών αποβλήτων. Χωρίς να θέλω να σταθώ περισσότερο στις κατά τα άλλα πολύ σωστές προτάσεις της ε, κυρίας Ρίπελ, θεωρώ ότι είναι ένα... Ε, συγγνώμη. Ε, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ... Ε, με, με ένα θέμα με διαστάσεις διεθνείς, ένα θέμα στο οποίο εμπλέκονται συμφέροντα διαφόρων ε, ισχυρών ρηπαντών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που όμως και εκείνη έχει ένα μερίδιο στην ε, ευθύνη και πρέπει να κάνουμε και εμείς την προσπάθειά μας για να περιορίσουμε τη ρήπανση ε, των θαλασσών και ακτών. Είναι καλή η πρόταση της Επιτροπής, ωστόσο παραμένουν κάποια σημεία αδύναμα ε, στα οποία θα πρέπει να σταθούμε και να τα διατυπώσουμε πιο ξεκάθαρους ε, όρους με βάση βέβαια τις προτάσεις της συντάκτηρας και τις φιλοδοξίες μας για την ευθύνη του παραγωγού, του κατασκευαστή καλύτερη θεωρώ ότι εδώ υπάρχει το εξής ε, πρόβλημα. Αφενός μεν ότι η διεύρυνση της ευθύνης του κατασκευαστή δεν ε, περιγράφει με ακρίβεια την έννοια του υπεύθυνου, του κυριολεκτικά υπέτειου της ρήπανση, γιατί η ρήπανση σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τη συμπεριφορά του ίδιου του καταναλωτή που δεν μπορεί να καταλογιστεί στον κατασκευαστή. Επίσης και το κόστος το οποίο αναφέρει και η κυρία Κάπλ. Δεν θα πρέπει να επιβαρύνουμε τους κατασκευαστές ε, κατά τρόπον ώστε τελικά να μετακυλήσουν αυτό το κόστος στον καταναλωτή. Ουσιαστικέ λύσει δεν έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, μια δεύτερη πτυχή ε, στην οποία εγώ εντοπίζω τα προβλήματα τα σχετικά με την, ε, με την ευθύνη του κατασκευαστή είναι ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό Ε, μια αγορά εδώ στην οποία τα προϊόντα αυτά μίας χρήσης είναι εισαγόμενα. Επομένως, ε, τα πλαστικά μίας χρήσης, επομένως ε, δεν υπάρχει δυνατότητα να φτάσουμε μέχρι τον κατασκευαστή, μέχρι τον αρχικό κατασκευαστή και να τον επιβαρύνουμε. Επιβαρύνουμε λοιπόν τον εισαγωγέα με την ευθύνη και το σχετικό κόστος. Ή επιβαρύνουμε μόνο τον εγχώριο κατασκευαστή χωρίς να μπορούμε αντίστοιχα να ελέγξουμε τον κατασκευαστή των ε, εισαγωμένων πλαστικών μίας χρήσης, τα οποία έχουν ακόμα, μεγαλύτερη, βέβαια, ε, ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο στη ρήπανση. Σε αυτό θα ήθελα κάποιες προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει κάνει μια προσπάθεια όχι όμως πιστική για μένα. Βέβαια και περιμένω και τις συζητήσεις με την συντάκτρια και τους ε, ισχυώδεις συγητές. Ευχαριστώ. Άλτε Βιάνικ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Κάπελ, αγαπητοί συνάδελφοι, χαιρετίζω την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώ ε, και το σχέδιο γνωμοδότηση των συναδέλφων μα από την ΕΝΒΗ. Τα τελευταία χρόνια καθίσατε λένε και σαφέστερο ο αντίκτυπο ε, του πλαστικού στο περιβάλλον μα. Η ευθύνη δεν βαρύνει μόνο του ε, τους κατασκευαστές ή τους καταναλωτές, μας βαρύνει όλους. Γι' αυτό οποιαδήποτε λύση θα πρέπει ε, να είναι διαρθρωτική, σφαιρική ε, και να αντικατοπτρίζει τις ε, ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. Πρέπει να μειώσουμε ξεκάθαρα και δραστικά την χρήση πλαστικών μίας χρήσης. Όμως αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Μόνο όταν υπάρχει βιώσιμη και οικονομικά προσιτή εναλλακτική λύση που είναι ουσιαστικά καλύτερη για το περιβάλλον. Και γι' αυτό στρεφόμαστε και προς τους επιστήμονες που εργάζονται άκουνα για να βρουν αυτές τις ε, βιώσιμες ε, εναλλακτικές λύσεις, τα υποκατάστατα. Και έτσι είναι πολύ σημαντικό ε, τα πλαστικά μιας χρήσης που καταναλώνονται ακόμα να ανακυκλώνονται. Και έτσι πρέπει να έχουμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ νομικών προποθέσεων και οικονομικών κινήτρων. Η πρόκληση του πλαστικού, από την άλλη, παρουσιάζει και πολλές ευκαιρίες. Επιπλέον χαιρετίζουμε ορισμένε από τι παρατηρήσει τη κυρία Κάπελ. Βλέπω ότι δίνει ευελιξία στα κράτη-μέλη να ελοποιήσουν τι πολιτικέ του με βάση τι ιδιαίτερότητε ε, τη ε, περιφερεια του. Όμω, ό,τι αφορά τι επισημάνσεις ή άλλες ε, απαιτήσει, πρέπει να διασφαλίσουμε την ομοιομορφία για λόγου αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και εύρυθμη λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Συνάδελφοι, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του πλαστικού και θα το πράξουμε. Ευχαριστώ. Äh, ναι, ευχαριστώ πολύ. Την ΚΟΕ θα ήθελα να ακούσω. Λόβε Περμέιο. Εσείς δεν μιλάτε εκ μέρους της ΚΟΕ. Ποιος ε, πρόκειται να λάβει το λόγο. Λόπες Περμέιο. Sí, estaba viendo sobre la opinión. Λοιπόν, για τη γνωμοδότηση, ε την κατάσταση για το μέλλον για την Ευρώπη. Ah, Όχι, αυτό είναι το επόμενο. Είμαστε ακόμα στα πλαστικά απόβλητα. Ναι, έτσι κατάλαβα. Συγγνώμη, συγγνώμη, αλλά κάποια στιγμή κάπου χάθηκα ε, και έκανα λάθος. Συγγνώμη. Καλώ, άρα δεν θέλει κανεί να λέει το λόγο του μέρου τη ΚΟΕ. Α και τα κάνουμε ένα μικρό ΑΕ, αν θέλει κανεί να παρέμβει. Όχι. Οι κυρίες μας εδώ είναι, έχουν ε, υπεροχή 6 προς 2 εντωμεταξύ ως προς την προσέλευση. Ξαναδίνω το λόγο στην συντάκτρια κυρία Κάπελ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους κοιόδης ε, συντάκτες. Βεβαίως συμφωνούμε ως προς την ουσία και την, ε, τη ματιά που ρίχνουμε στο πρόβλημα αυτό, την οπτική γωνία και το πρίσμα μας από το οποίο το βλέπουμε. Ε, είναι ένα διεθνές πρόβλημα, παγκόσμιο πρόβλημα. Ε, πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οπωσδήποτε ε, εναρμονισμένες προδιαγραφέ, μακάρι και στο παγκόσμιο επίπεδο για τις διευκρινήσεις σε σχέση με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάτι το οποίο θα μελετήσουμε ιδιαίτερα προσεκτικά στις συναντήσεις των σκιωδών ε, για την ευθύνη κυρίως του κατασκευαστή όπως υπόθηκε νωρίτερα. Προθεσμία πολύ σύντομη δυστυχώς για τις ε, τροπολογίες 6 Σεπτεμβρίου, γιατί 24 Σεπτεμβρίου, όπως μας είπε ο Πρόεδρος, έχουμε την ψηφοφορία για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την αντίστοιχη διαδικασία στην ΕΝΒΗ. Γίνεται όλο αυτό και βέβαια θα εντείνουμε και τις προσπάθειες σχέση με τους ε, συντονιστές για να είμαστε έτοιμοι στις 24 Σεπτεμβρίου για την ψηφοφορία. Σε ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ για την ε, διαθεσιμότητα να τηρήσετε και εσείς από πλευρά σας τις πολύ στενές αυτές προθεσμίες. Ο Πρόεδρος 24 Σεπτεμβρίου λέει ο Πρόεδρος τροπολογίες. Ξέρω ότι είναι διορθώνει ο Πρόεδρος, μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου τροπολογίες. Παρακαλώ όμως στα αγγλικά, δεδομένου ότι είναι τόσο στενές προθεσμίες μέχρι τις 24 που ψηφίζουμε και περνώ στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Εξέλιξη πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης με ένα σχέδιο γνωμοδότησης καθήλυν αρμόδια η ΑΦΚΟ, η Επιτροπή των Συνταγματικών Υποθέσεων. 21 Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου η ΑΦΚΟ έχει να ψηφίσει την εκθεσή τη. Εκ μέρου της Επιτροπής μας συντάκτρια είναι η συνάδελφος Μάλετιτ. που θα λάβει και το λόγο. Πέντε λεπτά παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Στην νομοδότηση χαιρετίζω την προσέγγιση που παρουσιάστηκε κατά την Ολομέλεια από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για το μέλλον της Ευρώπης. Από πλευράς οικονομικής πολιτικής, η γνωμοδότηση είναι μια ευκαιρία να επισημάνουμε και πάλι τη σημασία της ολοκλήρωσης διαδικασιών που ξεκίνησαν, ορισμένες τουλάχιστον, εδώ και χρόνια όπως η διαδικασία ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης και ε, η ανάγκη ε, να διασφαλίσουμε ένα ανοιχτό πνεύμα και ίση μεταχείριση όλων των ε, κρατών μελών ε, με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, μετά της Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών, με την ολοκλήρωση και εμβάθυνση της ΟΝΕ για την διατήρηση της ισορροπίας και της σταθερότητας μάλλον του ενιαίου νομίσματος, αλλά και της ευθυγράμμισης οικονομικών, δημοσιονομικών και εργασιακών πολιτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη-μέλη. Μας να επιπλέον πρέπει συνεχώς να έχουμε κατά νου ότι οι ε, επενδύσεις ε, και οι υπεύθυνε ε, οικονομικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις είναι βασικοί πυλώνες για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Εδώ αναφέρομαι και στο πρόγραμμα Invest EU, το οποίο είναι φρόζεκτο, θα αποτελέσει συνέχεια του ΕΦΣΥ και θα διασφαλίσει νέες επενδύσεις ε, που θα ε, φτάνουν ε, τα 30 δις ευρώ. Είναι σημαντικό να έχουμε μεγάλη έμφαση στην καινοτομία και στην κλιμάκωση των νεοφιών επιχειρήσεων. Έχουμε και το πρόγραμμα στήριξης διευθυντικών μεταρρυθμίσεων, γιατί ήταν πιλωτικό σχέδιο αρχικά. Ο αριθμός ετοιμάτων από τα κράτη-μέλη υπερεύει σε μεγάλο βαθμό τον αρχικό σχεδιασμό τα νέα προγράμματα μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να λάβουν την απαραίτητη στήριξη και στο νέο ΠΔΠ θα πρέπει να υπάρξει διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την εφαρμογή των ειδικών αναχώρα συστάσεων ε, στα κράτη-μέλη. Στην νομοδότηση θα πρέπει να τονίσουμε και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα ενιαίο φόρο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί εδώ και 25 χρόνια και έχει έρθει επιτέλους η ώρα να μειώσουμε το κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις, να περιορίσουμε τον κίνδυνο απάτης ΦΠΑ και να ενισχύσουμε ε, την εσωτερική αγορά και να ε, διευκολύνουμε το διασυνοριακό εμπόριο. Θα ήθελα εδώ να επισημανώ ότι εξεπλάγει όταν εξέτασα τη γνωμοδότηση της ΑΦΚΟ για το μέλλον της Ευρώπης, γιατί σε πολλά σημεία ε, στέκονται σε ζητήματα που άπτονται της ε, ΕΚΟΝ. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί. Ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία εδώ θα πρέπει να τα συζητούμε και εκεί να τα λαμβάνουν υπόψη. Και όχι όλα αυτά τα στοιχεία να επισέρχονται στην ε, γνωμοδότησή τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ιβάνα. Αντικαθιστά τον κύριο Μαυρίδη, κυρία Περές, εκ μέρους των Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για αυτή την παρουσίαση. Ο Κώστας Μαυρίδης μου ζήτησε να μιλήσω εξ ονόματός του. Ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα. Οι παρατηρήσεις που θα ήθελε να κάνει είναι αρκετές και αφορούν διάφορα θέματα. Κυρίως αφορά ότι όλη η προσέγγιση της Επιτροπής μας ε, στη συμβολή της, ε, στις εργασίες της ΑΦΚΟ θα πρέπει κυρίως να επικεντρωθεί πέραν των ε, πτυχών σε ποσοτικό επίπεδο, αλλά ε, να σταθεί και στα ποιοτικά κριτήρια και κυρίως ε, κοινωνικούς δείκτες ε, και πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό. Σε κάποια συγκεκριμένα σημεία θα ήθελε να προτείνει κάποιες τροπολογίες στην πρόταση της ηγήτριας, κυρίως για την Τραπεζική Ένωση. Ναι, μεν χαίρεται που υπάρχει μια ιδέα μιας ευέλικτης ασφάλειας, ε, ε, αλλά θα ήθελε να τεθεί το θέμα του έντις και της εγγύησης των καταθέσεων, να μην περάσει δηλαδή ε, χωρίς καμία παρατήρηση. Υπάρχουν πράγματα στα οποία μπορούμε να συμβάλλουμε εδώ στην Τραπεζική Ένωση. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, θεωρεί ότι υπάρχουν ε, προγράμματα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, το θέμα της ιδιοκτησίας, του ownership και ε, το να υπάρχουν ε, συστάσεις αναχώρα είναι κάποιες πτυχές τις οποίες πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω, κυρίως να λάβουμε υπόψη και την οικολογική μετάβαση και την δυνατότητα να συμπεριλάβουμε και κοινωνικά, ε, οικονομικά ε, και περιβαλλοντικά κριτήρια. Επίσης θεωρεί ότι ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να ενταχθεί στις ανησυχίες της Επιτροπής μας. Θεωρεί επίσης ότι στο θέμα της, ε, των οικονομικών και κοινωνικών αποκλήσεων στην Ευρωζώνη ε, θα πρέπει να έχουμε κάποια περαιτέρω στοιχεία, αρκετά στοιχεία και πάλι εδώ επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε ποιοτικά κριτήρια και τέλος όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής θεωρεί ότι οποιαδήποτε σχέση με την οικονομική διακυβέρνηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξεμήνου ε, θα έρθει σε αντίθεση με τους ίδιους τους στόχους ε, του Ταμείου Συνοχής. Αυτά λοιπόν τηλεγραφικά είναι τα όσα θα ήθελε να προσθέσει στις εργασίες. Ε, θεωρεί ότι το θέμα δεν είναι αμυγός οικονομικό, είναι ένα ε, πολύ σημαντικό πλαίσιο, διότι έρχεται και σε προεκλογική ε, περίοδο και ο καθένας θα πρέπει να πάρει θέση για να γνωρίζει και το όραμα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, αλλά και της Ευρώπης στο σύνολό τους, γιατί αυτά θα πρέπει να προτείνουμε και στις επόμενες ευρωεκλογές. Ευχαριστώ κύριε, Ευχαριστώ, κύριε Πέρας. Τσέλε. Αλντ ε, Λέ. Κορνίλια. Κορνίγη. Αλντε, παρακαλώ να πάρετε το λόγο. Ο κύριος Λούκη για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Ο ισκιώδης ηγητής, ο κύριος Τζίλε, ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να παρευρεθεί σε αυτή τη συνεδρίαση και θα διαβάσω τώρα μια δήλωση εκ μέρους του. Ο κύριος Ζήλε ευχαριστεί τον, ε, τη συντάκτρια της γνωμοδότησης, την κυρία Μάλετιτς, για τη δουλειά της και συμφωνεί ότι μεταξύ άλλων ε, η Ένωση των Κεφαλαιογορών θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπάρχουν μεταρρυθμίσεις ε, σε επίπεδο ευρωζώνης. Επίσης, ο κύριος Ζήλε θεωρεί ότι η γνωμοδότηση θα πρέπει να ανακλά περισσότερο την ομογένεια ε, στα θέματα αυτά. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να προωθήσουν την περαιτέρω ομοσπονδιακή πτυχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχουν και αρκετοί που είναι αντίθετοι. Και ακόμα και αυτοί που είναι κατά ε, την, ε, της περαιτέρω αδιαμφισβήτητης ομοσπονδιοποίησης της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουν να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε να συζητήσουμε λοιπόν πραγματικά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να συζητήσουμε και το γεγονός ότι συχνά υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις ε, πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Ζήλε θεωρεί ότι είναι απογοητευτικό ότι από όλε τις ιδέες ε, δεν αναφέρεται πουθενά όρο συνοχή, ενώ ταυτόχρονα στην έκθεση υπάρχουν κλήσεις για σύγκληση ε, για τις φορολογικές, εργατικές και οικονομικές πολιτικές. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε χωρίς να βελτιώσουμε το βιωτικό επίπεδο των νέων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, υπάρχει και η εμβάθυνση της ΟΝΕ. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι υπάρχουν ακόμα χώρε που δεν έχουν ευρώ και κάποιε από αυτέ κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ενταχθούν ποτέ στην ευρωζώνη. Η Ευρώπη του μέλλοντο ε, θα πρέπει να είναι μια Ευρώπη η οποία δέχεται του πάντε και όχι που δημιουργεί περαιτέρω έρηδε και κατηγορίε ε, και ε, μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Ο κύριο Ζήλιο προσβλέπει στι περαιτέρω συζητήσει και επικοδομητικές εργασίε. Ευχαριστώ. Κύριος Κορνία είναι εδώ για την Αλντε. Γκίγκολτ, πράσινη, επίση απουσίαζε. Και πάω στην ΚΟΕ. Κύριε το έχω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και η γενική έκθεση που παρουσίασε η Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων και η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας θα πρέπει να είναι στο ύψο των προκλήσεων δεν είναι μια τυχαία στιγμή για τη διαδικασία της ολοκλήρωσης και για το μέλλον μας. Το να συνεχίσουμε λοιπόν με μια λογική βάσει της οποίας ε, η καλύτερη λύση είναι περισσότερη Ευρώπη για όλα τα, τα δεινά τα οποία μας πλήττουν, σημαίνει ότι έχουμε χάσει ε, την προοπτική των όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Όσον αφορά τα θέματά μας, καταρχάς ε, ανησυχούμε βαθύτατα για τη γενικότερη αντίληψη που υπάρχει στην κατάρτιση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις αλλαγές που προτείνονται, όπως επίσης και στη μεταρρύθμιση των ίδιων πόρων το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιμείνει στην ιδέα ότι ο παρόν προπολογισμό είναι ανεπαρκή σαφέστατα για να ανταποκριθούμε στι ε, απαιτήσει ε, και στι ανάγκε ε, των Ευρωπαίων πολιτών. Επομένω, θα πρέπει να σταθούμε περισσότερο στι κοινωνικέ πτυχέ. Πέραν των όσων έχουν ανακοινωθεί και των δηλώσεων, ο προπολογισμό χάνει και τι δυνατότητέ του σε θέματα αλληλεγγύη και αναδιανομή και αυξάνεται σε θέματα τα οποία είναι καθαρά θέματα ασφαλείας. Θεωρούμε ότι θέματα όπως η Τραπεζική Ένωση ή η Ένωση κεφαλεγορών αξίζουν ε, πολύ πιο διεξοδική μελέτη. Δεν ε, ισχύει καμία Τραπεζική Ένωση και δεν είναι χρήσιμη καμία Ένωση κεφαλεγορών. Για να ολοκληρώσω, όσον αφορά την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η πρόταση να ολοκληρώσουμε και να αυξήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτή το ρόλο του ευρώ δεν μπορεί να παραβλέψει και την όλη συζήτηση όσον αφορά τι ελλείψει του σχεδιασμού του ίδιου του ευρώ. Για να μπορέσουμε να έχουμε μηχανισμού για να απαντήσουμε στα ασύμετρα ε, σοκ τα οποία θα συνεχίσουν να ε, εμφανίζονται συνεχώς και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το πόσο κακή ήταν η διαχείριση της ε, οικονομικής κρίσης, διότι αυξήθηκαν οι αποκλήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι αποκλήσει εντός των ίδιων των χωρών. Υπάρχουν αρκετοί πολίτες που ανησυχούν ε, για τις συνέπειες της αύξησης των ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς δεν μπορούμε να λέμε ότι η ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης είναι καλή ιδέα, χωρίς να αναρωτηθούμε και τι συνέπειες έχει το παρόν μοντέλο και τι ε, ε συνέπειες είχε για όλα τα δυνάτα τα οποία μας πλήττουν αυτή τη στιγμή. Η προϋπόθεση λοιπόν για να είναι χρήσιμη αυτή η διαδικασία για τους πολίτες μας σημαίνει ότι θα πρέπει να θέσουμε και τα κατάλληλα ερωτήματα. Καταρχάς, οι παλιές συνταγές ε, που εφαρμόζοντας ε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αποτελούν τμήμα του προβλήματος και επομένως χρειαζόμαστε νέες λύσεις για να επιλύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η FTD και μόνο. Θέλετε το λόγο κύριε Μόνο. Όχι, καλώς. Ενφ, όχι, δεν άλλος κανείς παρόν εδώ. Και άρα Άι, εάν θέλει κανείς το λόγο. Όχι. Εσείς, κυρία συνάδελφε, θέλετε για να κλείσουμε να πάρετε πάλι το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, για τη συμβολή τους σε αυτή τη συζήτηση και θα ήθελα να τονίσω ότι επειδή υπάρχει ε, και περιορισμός χώρου, ε, τονίσαμε απλώ κάποια γενικά στοιχεία στη γνωμοδότηση και τις επόμενες εβδομάδες ε, σίγουρα θα μπορέσουμε να προσθέσουμε και κάποια πράγματα τα οποία απουσιάζουν και να τονίσουμε και κάποια σημαντικά στοιχεία στη γνωμοδότηση. Επίσης, αναφέρθηκε επίσης ότι δεν λέμε περισσότερα για το έντις και την εγγύηση των καταθέσεων και τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων και τις οικονομικές και κοινωνικές αποκλήσεις και επίσης τη συνοχή και τη σύγκληση. Αυτά σίγουρα είναι στοιχεία τα οποία θα ε, συμπεριλάβουμε στις επόμενες εβδομάδες και θα ήθελα να πω ως μέλος και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ότι ασχολούμαστε εκεί ε, πολύ επισταμένα με τα θέματα της συνοχής. Γι' αυτό λοιπόν δεν θεώρησα εδώ, σε αυτή τη γνωμοδότηση, ότι πρέπει να έχουμε κάτι συγκεκριμένο γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ και από πλευράς μου τελευταία σχόλια. 12 Σεπτεμβρίου τροπολογίες, 5 Νοεμβρίου συζήτηση και ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης κοινό σύστημα ΦΠΑ σε σχέση με ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες που είναι εκτιθμένα στην απάτη και φοροαποφυγή ΦΠΑ. Σχέδιο έκθεσης Πρώτη εξέταση. Κυρία είναι. Ο κύριος Πιετικάιν δεν είναι εδώ όμως σήμερα. Τον αντικαθιστά όμως. Την αντικαθιστά. Διορθώνει ο πρόεδρος και μας παρουσιάζει το θέμα αυτό που ε, παρουσιάζεται από το άρθρο 50, στην απλοποιημένη διαδικασία, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ε, προβλήματα. Το σχέδιο έχει κατεθεί στις 17 Ιουλίου. Η προθεσμία για την κατάθεση αντιρρήσεων είναι δεκαήμερη κανονικά, με παράταση έως την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, λέει ο Πρόεδρος. Ε, Αλλιώς πάμε για την πρώτη ολομέλεια του Οκτωβρίου με την απλουστευμένη διαδικασία. Η τοποθέτηση τώρα της κυρίας Πιέτη και σας τη διαβάζω. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε δει το σχέδιο εκθέσεως ε, για ε, οδηγία του Συμβουλίου για ένα μηχανισμό ταχείας αντίδρασης κατά της φοροαποφυγής ΦΠΑ. Στόχο έχουμε την παράταση καταρχάς, την επέκταση του δυνατότητα για τα κράτη-μέλη για την επέκταση του κανονισμού αρχαίας αντίδρασης με βάση και την οδηγία και το μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης σε περιπτώσεις μαζικής απάτης. Μέτρα χρήσιμα για τα κράτη-μέλη ως στοχευμένα και προσωρινά εκπνέουν όμως στις 31 Δεκεμβρίου του 2018. Η παράτασή τους μέχρι τον, τα Ιουνίου του 2022 επιτρέπει στα κράτη-μέλη την αξιοποίηση των αποτελεσματικών αυτών εργαλείων και την αντιμετώπιση ευνίδιων μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων απάτης. δεδομένου ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και δεν προκύπτουν συνέπειες αρνητικές για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα ε, δεν γίνανε πολιτικά ζητήματα ε, το θέμα αυτό. Προτείνω, μας λέει η κυρία Πιερτικάινεν, να ακολουθήσουμε τις προτάσεις με βάση βέβαια και τον περιορισμένο χρόνο και τους πόρους του περιορισμένου της Επιτροπής μας. Η κυρία Πιερτικάινεν λοιπόν προτείνει να ακολουθήσουμε τις, τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευχαριστώντας μας για τη συνεργασία. Uh, of um, uh, And uh, Αυτά μας λέει η εισηγήτρια που δεν είναι εισηγητής και δίνω το λόγο στους Σκιώδης. Σοσιαλιστές δεν έχω. Έχω. Υπέρ Πέρες. Μάλιστα. Οι σκιώδες μας ζητά συγγνώμη που δεν βρίσκατε εδώ σήμερα. Ο κύριος Καγνιγέ. Ε, Συμμερίζεται σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις της εισηγήτριας, εφόσον πρόκειται και για τεχνικές προτάσεις υπάρχει αυτός ο μηχανισμός ε, της αντιστροφής της επιβάρυνσης, ελήψη ενός ε, συνολικού πλαισίου για τον ΦΠΑ που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να το χρησιμοποιούν για την καταπολέμηση της απάτης ΦΠΑ ε, το να μπορούμε να συνεχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε αυτό το σύστημα μέχρι το 2022 είναι κάτι το οποίο μπορούμε να δεχτούμε. Και έτσι δεν θα φέρουμε αντίθεση και αντίρρηση στην ταχεία διαδικασία έγκριση τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμω, επί τη ευκαιρία, μπορούμε να υπενθυμίσουμε ότι για τη δική μα πολιτική ομάδα η επεξεργασία, οριστικοποίηση, διαπραγμάτευση και θέση σε ισχύ ενό ε, ολοκληρωμένου συστήματος ΦΠΑ είναι επίγουσα σημασία ε, και το, είναι κάτι το οποίο αναφέρουμε καθ' όλη τη διάρκεια τη θητεία αυτή. Ευχαριστούμε πολύ, Πεβάνς. Η Case Winburn είναι στο καταλογό μου πλευρά ε, στηρητικών μεταρρυθμιστών. Δεν βρίσκεται κάποιο εδώ όμω, ούτε σκιώδη ε, υπάρχει. Α! Η Λίβε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος του κυρίου Κογνιγέ, που είναι σκιώδης για αυτό το φάκελο, να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Πιατικάινεν, την εισηγήτρια. Η Άλντε θα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για να έχουμε ε, συγκεκριμένη ε, πρόοδο και επιτάχυνση της νομοθετικής διαδικασίας. Εδώ και πολύ καιρό μιλούμε για την Ένωση των Κεφαλαιογορών. Στι επόμενε εβδομάδε, ο κύριος Κογνιγέ με τα χαρά ε, θα συνεργαστεί με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, Λίβε. Πράσινη. Κάτω, σκιώδης δεν είναι κανείς εδώ όμω να την, να την εκπροσωπήσει υποψιάζει. Γκουε το ίδιο, η FTT, Μονρό. Μονό, κύριε Μονό. No, thank you κύριε Πρόεδρε. Ενφ, ουδής, διάει κανείς, δεν ενδιαφέρεται και έτσι σας ενημερώνω. ότι η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών εκπνέει στι 6. Πρώτη ολομέλεια του Οκτωβρίου θα συζητήσει το θέμα. Περιμένουμε τις περαιτέρω συζητήσεις μαζί σας. Και μπορώ να περάσω ευθέω στο σημείο 6 από το ενδεικτικό και τονίζω ενδεικτικό είναι πάντα χρονοδιάγραμμα προβλέπεται για τις 4 ε, το θέμα αυτό και έτσι δεν έχω ούτε τον εισηγητή ούτε και τους περισσότερους σκιώδεις που θα έπρεπε να είναι εδώ και διακόπτω μέχρι τις, 6, μέχρι τις 4.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

So, dear colleagues, um, as agreed, it's 4 p.m. We... Ε, μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι την Επιτροπή τη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών και Επιστηματικών Υποθέσεων σημείο 6 Γνωστοποίηση σχετικά με τις αηφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας και τροποποίηση της οδηγίας σχέδιο γνωμοδότησης ΕΜΠΛ Envy Farm, γνωμοδότηση. Ο Πολ έχει την έκθεση και το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν ξεκινήσαμε τη θητή αυτή, το συζητούσαμε την ε, αγαπητή συντονίστρια, υπήρχε μια πρόταση για μια ένωση των κεφαλαγορών. Όμως, δεν υπήρχε καμία συζήτηση για τη βιωσιμότητα. Τώρα όμως έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και θεωρώ ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε σημαντικό ρόλο εδώ και με την ε, τροποποίηση της νομοθεσίας αλλά και ασκώντας πίεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς άλλους ε, για να αναδειχθεί το ζήτημα. Το Ηνωμένο Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει ε, μία έκθεση πρωτοβουλίας, ε, με καθυστέρηση βέβαια, αλλά εξακολουθεί να είναι χρήσιμη. Γιατί η πρόταση που συζητούμε σήμερα έχει ήδη συζητηθεί υπό τη μορφή έκθεσης πρωτοβουλίας. Το Κοινοβούλιο λοιπόν με ευρεία πλειοψηφία είπε ότι θέλει να υπάρχει υποχρεωτικό ε, πλαίσιο δεσμευτικό πλαίσιο που να λαμβάνει υπόψη τις ε, αρχές ε, του UNPRI αλλά ε, και τις κριτήρες γραμμές του ΟΣΑ του 2017. Η νομοθεσία που έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης ήταν πιο μετριοπαθές, ενώ ο αρχικός στόχος ήταν να δώσουμε έμφαση και στις υποχρεώσεις των επενδυτών που πρέπει να λάβουν υπόψη και τους μη χρηματοοικονομικούς παράγοντες και ουσιαστικά τι πρόκειται για τη δέωσα επιμέλεια. Τι λέει λοιπόν αυτή η έκθεση ότι χρειαζόμαστε, ξέρουμε μάλλον πώς λειτουργεί η δέωσα επιμέλεια και θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τους επενδυτές. Γιατί πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ε, ο χρηματοοικονομικός παράγοντας και ο μη χρηματοοικονομικός παράγοντας. Πρόκειται λοιπόν για μία τροποποίηση και ο στόχος του Κοινοβουλίου είναι μια αλλαγή νοοτροπίας των επενδυτών. Ότι δηλαδή δεν πρέπει να σας απασχολούν μόνο τα χρήματα, αλλά να έχετε ένα ευρύτερο και πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Και χρονικά. Αυτή είναι η ουσία της ε, έκθεσης. Στην τροπολογία 13 επίσης αναφέρεται ότι δεν θα πρέπει ε, η γνωστοποίηση ή η η επιμέλεια να αφορά μόνο ε, τον αντίκτυπο βιωσιμότητας των επενδύσεων, αλλά να αφορά όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, είτε, πρόκειται, είτε υπάρχει στόχευση είτε όχι. Βεβαίω, επιμέλεια λοιπόν όπως έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και πάλι δεν είναι μόνο για τις πράσινες επενδύσει, αλλά για όλες τις επενδύσει. Και ένα άλλο στοιχείο είναι ότι όλοι ξέρουμε ότι σημαντική, σημαντικός διάβλος χρηματοδότησης είναι ο τραπεζικός κλάδος. Όχι μόνο τα στεξιοδοτικά ε, οι διαχειριστέ περιουσιακών στοιχείων, οι ασφαλιστικέ, αλλά και άλλοι φορεί. Έχουμε συμπεριλάβει την ε, αηφορία εδώ και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί και ο τραπεζικός κλάδος ε, είναι ευάλωτος ε, σε τέτοιους κινδύνους που αφορούν τη βιωσιμότητα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ ε, ασφαλιστικών, συνταξιδοτικών ταμείων αφενός και τραπεζών αφετέρου. Γι' αυτό θέλαμε να συμπεριλάβουμε τον τραπεζικό κλάδο εδώ, με την ε, τροπολογία 13. Μετά, στην έκθεση πρωτοβουλίας, είχαμε πει ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε την οτροπία, που είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να ακολουθούμε και το δίδαγμά μας. Επομένω, όπως λέμε και στην τροπολογία 13, θα πρέπει η αποζημίωση να αφορά και τους ε, μη χρηματοοικονομικούς παράγοντες και να συνδέεται με την ε, βιωσιμότητα. Και αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με, την, ε, με το πρασίνισμα της οικονομία. αφορά και κοινωνικού παράγοντε. παραβίαση ανθρωπινών δικαιωμάτων, υφαρπαγή γη, τα οποία δεν τυποποιούνται εύκολα, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και φυσικά ζητήματα διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένη και τη ε, φόρου αποφυγή. Τέλο Πρόεδρε. Στην IORP συζητήσαμε το ζήτημα των κατεξουδότηση πράξεων. Από τη συζήτηση θυμάμαι ότι υπήρχε ιδιαίτερη αντίσταση στην ε, συμπερίληψη των κατεξοδότηση πράξεων εδώ. Θεωρήσαμε ότι δεν ήταν πολύ παραγωγική και γόνιμη στάση και ότι έπρεπε να αλλάξουμε. Αντί να έχουμε κατεξοδότηση πράξης, προσθέσαμε ή προσπαθήσαμε να προσθέσουμε απευθείας ε, στην οδηγία τα ζητήματα ε, του Ιδρύματος Επαγγελματικών Συνταξιωτικών Παροχών IORP. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτές ήταν ε, οι κύριες αλλαγές σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής, αλλά ελπίζω το έργο μας να προχωρήσει γρήγορα για να ολοκληρωθεί εντός της θητείας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Πολ. Εξ ονόματος της ε, σκιώδους ηγήτριας κυρίας Πιέτη Κάινεν, το λόγο έχει η κυρία Μάλετιτς. Ευχαριστώ πολύ. Θα διαβάσω μόνο τη δήλωση της συναδέλφου. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για τα όσα έχει κάνει, για αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση. Σήμερα ξεκινούμε ε, τη συζήτηση ε, για την, την πρώτη νομοθετική πρόταση της ευρύτερης δέσμης για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά. Ε, που είναι ένα απαραίτητο βήμα λαμβάνοντα υπόψη και τις συστάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκε τον Μάιο. Αυτή η πρωτοβουλία είναι πραγματικά ρεζοσπαστική γιατί θέλουμε να μετριάσουμε και τον ε, οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των επενδύσεων. Θέλουμε να στραφούμε προς επενδύσεις με χρηστές διαδικασίες ο κίνδυνος ε, βιωσιμότητας και η επιθυμία μετριασμού του κινδύνου βιωσιμότητας είναι ε, κάτι το ρεαλιστικό και το ευπρόσδεκτο. Βλέπουμε ότι αυξάνεται αυτός ο κίνδυνος και αν δεν ε, μεριμνήσουμε για τον μετριασμό του μπορεί να θέσει ένα αμφιβόλο την οικονομική σταθερότητα. Πρέπει λοιπόν ε, να διασφαλίσουμε ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά λαμβάνουν επαρκώς υπόψη αυτόν τον κίνδυνο και στις επενδυτικές τους αποφάσεις. Και έτσι μπορούμε ε, να δώσουμε τα σωστά κίνητρα στους συμμετέχοντες στην αγορά και να αποθαρρύνουμε ε, τη μη λελογισμένη λήψη αποφάσεων. Και οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν λογογνώσεις και εδώ είναι σημαντικές ε, οι δημοσιεύσεις αυτές, οι γνωστοποιήσεις, γιατί έτσι μπορούν οι συμμετέχοντες στην αγορά να έχουν ε, επαρκείς πληροφορίες για τον αντίκτυπο στη βιωσιμότητα. Επομένως, η υποχρέωση γνωστοποίησης θα πρέπει από κοινού και πλέραν των επενδυτών μάλλον να καλύπτει και έναν ευρύτερο κατάλογο επιχειρήσεων και το καθεξής στις οποίες γίνονται οι επενδύσεις. Η πρόταση ε, του πακέτου βιώσιμων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι κάτι το απαραίτητο για τη μετατόπιση των χρηματοοικονομικών ροών προς τη στήριξη τη οικονομία χαμηλή κατανάλωσης άνθρακα και προκειμένου οι αποζημιώσεις μας, ε, συγγνώμη, οι αποταμιεύσει μα θα είναι εξασφαλισμένε σε επόμενε δεκαετίες και ότι θα έχουμε επενδύσει σε υποδομέ. Ε, που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν και τις ε, προεκτάσεις κλιματικής αλλαγής. Αντίστοιχα, πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα με το μέγεθος ε, του οργανισμού και με τον κίνδυνο της ε, εν λόγω δραστηριότητας και να υπάρχει επιμερισμός του κινδύνου και του άχθους, ιδίως για τις μικροσές επιχειρήσεις. Τα μέτρα ε, θα πρέπει λοιπόν να εφαρμοστούν και με αναλογικό και μεταβατικό τρόπο. Προβλέπω συνεργασία με τον εισηγητή και τους χειώδες. Ευχαριστούμε. Εξ ονόματος ε, του συναδέλφου Καμάλ, Ζανταλούς για το ECR. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Ε, αντικαθιστώ τον Σαγίτ που ζητά συγγνώμη, θέλει να εργαστεί για αυτό το φάκελο στο μέλλον και μου ζήτησε να διαβάσω τη δήλωσή του. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε φυσικά και τον εισηγητή. Σε ό,τι αφορά τις βιώσιμες και υπεύθυνε επενδύσεις είναι πολύ θετικό που βλέπουμε ότι το σύνολο του κλάδου σημειώνει σημαντική πρόοδο ε, σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική και οικονομική υπευθυνότητα είναι πλέον ένα σημαντικό κριτήριο για τις επενδυτικές αποφάσεις και στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο και αυτό είναι πολύ θετικό. Σε ό,τι αφορά τώρα πιο συγκεκριμένα το σχέδιο γνωμοδότηση ε, του κυρίου Τάγκ, ε, λέει ο Καμάλ ότι πρέπει να έχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ βιώσιμων επενδύσεων, αλλά και να μην έχουμε μία και μόνο λύση για όλους. Υπάρχει μία σειρά παραγόντων που πρέπει να λάβουν υπόψη προκειμένου οι επενδυτές να είναι σε θέση να πάρουν τις σωστές αποφάσεις έχοντας ε, πλήρη εικόνα της κατάστασης στην αγορά. Πρέπει να έχουμε κατά νου και την ε, πολυμορφία των ε, κλάδων που εμπίπτουν στο πεδίο αυτής της νομοδότησης από συνταξιδοτικά ταμεία και το καθεξής. Πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη ευελιξία κατά την εφαρμογή και να δίνουμε παράλληλα πρόσβαση στους επενδυτές στην πληροφορία για λόγους δέους επιμέλειας. Ο Σαγίτ Καμάλ επίσης ε, με τα χαράσεις βλέπει ότι ο εισηγητής ε, αναφέρεται στη βιωσιμότητα σε σχέση με ε, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και την κοινωνική ευθύνη και βιωσιμότητα και να διευρύνουμε το σημείο εστιασή μας. Γιατί έχουμε μια πιο σφαιρική ε, προσέγγιση ως προς τη βιωσιμότητα και μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε ευρύτερα ζητήματα όπως η ανέχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός ε, και οι επιζήμιες επενδυτικές πρακτικές. Αλλά σίγουρα θα ε, καταλήξετε σε σωστές προτάσεις από κοινού ε, χαιρετίζει τη συμπερίληψη του τραπεζικού κλάδου στην πρόταση του συγητή. Είναι σημαντικό ε, και οι τράπεζε να αποδίδουν τη δέουσα σημασία ε, στους παράγοντες ESG. Έχουμε δει και στο παρελθόν από ε, προηγούμενες ε, νομοθετικές προτάσεις ότι υπάρχουν θεμελιώδεις ε, αλλαγές μεταξύ πιστοτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών ιδρυμάτων. Γι' αυτό και υπάρχει και ξεχωριστή νομοθετική μέρημνα. Μπορεί λοιπόν να δημιουργεί πρόβλημα εδώ με τη συμπερίληψη του τερβαζικού κλάδου, αλλά θα δούμε ανάλογα και με την προσέγγιση που θα ακολουθήσει ο εισηγητή. Ω ECR θέλουμε το τελικό αποτέλεσμα να επιτρέπει ε, στους επενδυτές να παίρνουν τις αποφάσεις ε, έχοντας πλήρη εικόνα της κατάστασης Ξέρουμε ότι πολλά μένουν να γίνουν, αλλά προβλέπουμε στη συνέχεια τη συνεργασία με τον εισηγητή και του κοιόδη για να έχουμε ένα πολύ επικοδομητικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Λίβη ήταν εδώ εκ μέρου τη Άλντε, Λίβε Βίρινγκ, αλλά δεν είναι εδώ πια. Κύριος Γκίγκολτ, λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Εκ μέρου τη κυρία Σκοτ Κάτω. Όντω, Πρόεδρε, αγαπητέ Ζήμων. Έχω στα αγγλικά τις ε, σημειώσεις της Μόλι. Θα μπορούσαμε να έχουμε περιοριστεί σε ένα έβγε Πολ. Αυτό θα έλεγα εγώ. Αλλά δεν μου ζήτησε η κυρία Σκοτ Κάτω να σου πω μόνο έβγε. Θα σου διαβάσω λοιπόν το εξή. Οι προσπάθειε του συντονιστή για να ολοκληρώσουν τι διαδικασίε για την ε, αποκάλυψη των ε, ε, συμμετεχόντων στην αγορά οδηγεί σε ένα καθεστώς με πληροφορίες ε, σημαντικές για τον επενδυτή που εξασφαλίζουν ταυτόχρονα ότι οι παρέχοντες της ε, επενδυτικής υπηρεσίες θα μεριμνούν έτσι ώστε να ενημερώνουν κατάλληλα θετικέ αλλαγές που μας προσφέρει στην πρόταση επιτροπή σε αυτό το σχέδιο είναι η εισαγωγή του κινδύνου βιώσιμότητα, η εισαγωγή της έννοιας της βιώσιμης επένδυσης. Ιδιαίτερο ευπρόζεκτο είναι το γεγονός ότι το σχέδιο έκθεσης προσπαθεί να περιγράψει τους κινδύνους για τον επενδυτή και όχι μόνο για την απόδοση. Περιλαμβάνει απεριόριστα, ε, απερίφραστα τις ε, τράπεζες και ορίζει ότι θα πρέπει οι πολιτικές να αποφεύγουν βέβαια και την επιβάρυνση της βιωσιμότητας αλλά ταυτόχρονα και να δίνουν κίνητρα για ενίσχυση αυτής. Θα συνεργαστούμε με τον συντάκτη, με τον εισηγητή για καλύτερες τροπολογίες. Με χαρά λοιπόν ελπίζω να το απέλαυσες, να το απόλαυσες Πολ και στο παραδίδω. Ευχαριστώ. Μακάρθι Γκούε θα έπρεπε να είναι εδώ, αλλά δεν είναι. Κύριε Μονό, πάλι εσείς. Θέλετε το λόγο όχι και πάμε στο ΙΕΝΕΦ που δεν θέλει το λόγο. Ο κύριος Στάν. Πολύ γρήγορα προχωρήσαμε έτσι και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που ήρθαν εδώ και διάβασαν τα κείμενά τους. Ευχαριστώ πολύ. Το εκτιμώ που έστω κάνατε τον κόπο. Να πω σύντομα ότι σε αυτό το στάδιο της συζήτησης ε, προσβλέπω σε επικοδομητικές συζητήσεις. Νομίζω ότι ήδη έγινε διεξοδική και αναλυτική ε, συζήτηση για αυτή την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας που σημαίνει ότι περιλαμβάνει όχι μόνο την βιωσιμότητα υπό την έννοια την οικολογική αλλά και ε, την χρηστή διακυβέρνηση και συμφωνώ και με τη Σύρπα ότι πρόκειται για μια πολύ καινοτόμα πρωτοβουλία. Αυτό πρέπει να γίνει προκειμένου ο χρηματοπιστωτικός τομέας να αλλάξει και να στραφεί προς τη βιωσιμότητα με την ευρεία τη έννοια. Αυτό, κατά την άποψή μου, περιλαμβάνει και τις τράπεζες. Είναι πολύ σημαντικός διάβλος, δεν μπορούμε να τον παραβλέψουμε και ε, είναι τελείω διαφορετική μεταχείριση, για παράδειγμα, για τα σταξιοδοτικά ταμεία και τις τράπεζες. Ε, αλλά από την άλλη, πρέπει πάντα να εξετάζουμε και το στοιχείο της αναλογικότητα. Ε, και δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια λύση πανάκια για τα πάντα. Αυτό λοιπόν είναι το άνοιγμα που έχουμε σε αυτή τη συζήτηση και θα ήθελα να έχουμε μια γενική προσέγγιση η οποία θα στοχεύει προς συγκεκριμένους παράγοντες για κάθε προϊόν και για κάθε παραγωγό αλλά ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίζουμε δεν θα είναι ο ίδιος για κάθε παραγωγό και για κάθε προϊόν. Θα είμαι σύντομος λοιπόν κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστώ τους πάντες για την συμβολή τους και προσβλέπω στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Από πλευρά μόνο προθεσμίες 5 Σεπτεμβρίου για τις τροπολογίες 18 Οκτωβρίου συζήτηση 5 Νοεμβρίου ψηφοφορία. Σημείο 7 τώρα της κυρίας Δελάνγκε και Γκαλτιέρη, Γκουαλτιέρη που δεν είναι εδώ κύριος Γκουαλτιέρη στις 4.30 μπορεί να έρθει. Άλλη μια φορά λοιπόν διακόπτουμε για να συνεχίσουμε στις 4.30.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

Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τις εργασίες μας και πάμε στα... στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης το οποίο γνωρίζετε είναι μια κοινή συζήτηση για τις δύο νομοθετικές προτάσεις του πακέτου NPF ο κανονισμός ε, για την ελάχιστη κάλυψη απολειών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ε, οι ε, αγορές ε, πιστώσεων, οι υπηρεσίες πιστώσεων και η ανάκτηση των εγγύσεων. Όπως γνωρίζετε έχουμε δύο συνεισηγητές, εγώ είμαι ένας εκ των συνεισηγητών και η άλλη είναι η Στέρντε Λάγκε. Επομένως είναι μια καλή ευκαιρία να τα συζητήσουμε μεταξύ μας ε, και μεταξύ των συνεισηγητών, γιατί είχαμε και τις καλοκαιρινέ διακοπές, επομένως ε, δεν μας δόθηκε ευκαιρία να συζητήσουμε και πάρα πολύ. Θα είναι μια πολύ ανοιχτή πρώτη ε, ανταλλαγή απόψεων. Οι συνεισηγητές έχουν 8 λεπτά ο καθής. Εστέρ, θέλει να ξεκινήσεις. Ναι, βεβαίω. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που είναι παρόντες εδώ, διότι πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η συζήτηση είναι ένα θέμα το οποίο όπως γνωρίζετε όλοι σας ε, ήταν ήδη στην ε, ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2015 για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Αναφέρθηκε το θέμα της, ε, του επιμερισμού του κινδύνου και υπάρχουν και δύο κρεμότητες λοιπόν ακόμα από την ανακοίνωση αυτή όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου. Το ένα είναι η... Ε, μεταχείριση των τραπεζών για την έκθεση ε, σε κάποιους κινδύνους και το άλλο είναι η έκθεση σε μη εξυπηρετούμενες ε, πιστώσεις, που είναι αυτό που συζητάμε τώρα. Και έχουμε δύο προτάσεις, έχουμε και τον κανονισμό και την οδηγία. Εγώ θα επικεντρωθώ στο πρώτο και έχω ελάχιστες παρατηρήσεις για την οδηγία. Για τον κανονισμό, που στόχο έχει να περιλάβει διατάξεις που αφορούν την μείωση των κονδυλίων των τραπεζών εάν δεν καλύπτονται επαρκώς ε, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Εδώ ε, περιμένω να ακούσω διάφορες απόψεις σήμερα. Οι συνεισηγητές ε, αντέλεξαν απόψεις ε, για τα θέματα αυτά πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά υπάρχουν θέματα στα οποία ακόμα πρέπει να βρούμε κοινό έδαφος, επομένως ε, καλό είναι να ακούσουμε και τους συναδέλφους. Θα σας κάνω μια παρουσίαση των βασικών στοιχείων που έχουμε λοιπόν. Πρώτον, η αναλογία της έκθεσης που θα πρέπει να καλύψουμε. Θα πρέπει να αυξάνεται χρονικά, δηλαδή πιο πολύ προς το τέλος του χρονικού περιθωρίου ή να είναι γραμμική αύξηση. Και μπορεί πράγματι όσο μεγαλύτερη είναι μια εξυπηρέτηση της έκθεσης, ε, τόσο πιο δύσκολο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι να αποπληρωθεί ε, στο τέλος ε, ή θα μπορούσε να πει ότι αφού το βλέπεις το πρόβλημα γιατί δεν το αντιμετωπίζεις ευθύ εξ αρχής και να αρχίσεις να έχουμε τουλάχιστον μια γραμμική προσέγγιση γιατί να περιμένουμε δηλαδή μέχρι να διωγγωθεί το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο είναι κατά πόσο γίνεται διάκριση μεταξύ των λόγων για τους οποίους ε, δεν έχουμε εξυπηρέτηση της έκθεσης αυτής. Δηλαδή, κάνουμε διάκριση μεταξύ αυτών που έχουν καθυστέρηση πάνω των 90 ημερών ή δεν υπάρχει καμία εξυπηρέτηση για άλλους λόγους. Εγώ ειλικρινά δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε σαφή διάκριση μεταξύ των δύο. Διότι ορισμένες φορές ε, έκθεση για την οποία δεν υπάρχει εξυπηρέτηση ε, μπορεί για πολλούς λόγους να μην αποπληρωθεί καθόλου, ακόμα και ε, για περιπτώσεις οποίες έχουμε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Ε, υπάρχει βέβαια και η διάκριση μεταξύ ασφαλισμένων και μη ασφαλισμένων ε, δανείων. Ε, η Επιτροπή λέει ότι πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ αυτών και των άλλων αλλά και συμφωνούν όλοι, αλλά υπάρχει διάσταση απόψεων να αφορά το επίπεδο φιλοδοξίας σε αυτές τις δύο ομάδες ε, μη εξυπηρέτηση. Όσον αφορά τον αριθμό των ετών που προσφέρονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος, εδώ έχουμε διάφορες απόψεις μεταξύ 2 και 5 ετών για τα μη ασφαλισμένα ε, μη εξυπηρετούμενο και 7 έως 12 για τα ασφαλισμένα. Ε, και υπάρχει και το θέμα του επίπεδου της συνολικής κάλυψης. 100% κάλυψη και στις δύο περιπτώσεις, και για τα ασφαλισμένα και τα μη ασφαλισμένα. Γίνεται διάκριση ε, λιγότερο για τα ασφαλισμένα. Προτείνεται ένα φάσμα μεταξύ 70% και 100% το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Ένα άλλο θέμα είναι κατά πόσον θα κάνουν και άλλες διακρίσεις ε, στην όλη συζήτηση. Παραδείγματο χάρη, διάκριση μεταξύ ε, του επίπεδου της ανησυχίας ή το κατά πόσον ε, έχει γίνει ανεξάρτητη αξιολόγηση ή διάκριση μεταξύ βιώσιμων και μη βιώσιμος, ε, βιώσιμων μέτρων αντιμετώπισης. Εγώ πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον μια τράπεζας να επιτρέψει μόνο βιώσιμα μέτρα. Τώρα το κατά πόσο να αυτή η διάκριση ε, προσωπικά αμφιβάλλω. Για το ΕΛΚ όπως και να έχει πρέπει να υπάρχει ένα δίκαιο σύστημα. Δηλαδή θα κάνουμε διάκριση στο επίπεδο της φιλοδοξίας και στην ταχύτητα μεταξύ των ασφαλισμένων και μη ασφαλισμένων, ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά πρέπει κάπως να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Προς το παρόν αυτά τα οποία βάζουμε στο ε, τραπέζι είναι η διάκριση μεταξύ των δύο κατηγοριών. Η Κομισιόν κάνει διάκριση μεταξύ τεσσάρων κατηγοριών και υπάρχει και η ιδέα, εάν προσθεθούν επιπλέον κριτήρια, να φτάσουμε σε 8 διαφορετικές κατηγορίες έκθεσης λόγω μη εξυπηρετούμενων δανείων. ασφαλισμένα, μη ασφαλισμένα, ασφαλισμένα με ανεξάρτητη αξιολόγηση, απλώς ασφαλισμένα κλπ. κλπ. Δεν ξέρω αν περιπλέξουμε περαιτέρω μια τόσο δύσκολη πρόταση ε, θα καταφέρουμε τίποτα. Ε, το θέμα είναι πόσες μεταβλητές θα συμπεριλάβουμε ε, και αυτό πρέπει να συζητηθεί και φυσικά το πεδίο εφαρμογή είναι κάτι τελευταίο. Η Επιτροπή λέει ότι θα καλύψουμε την έκθεση μόνο σε περίπτωση που δημιουργηθεί μετά από την ημερομηνία της πρότασης. 14 Μαρτίου του τρέχοντος π.χ. Αυτό σημαίνει ότι θα παραβλέψουμε όχι μόνο δάνεια τα οποία αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετούνται, αλλά και δάνεια τα οποία υπάρχουν και μπορεί να αρχίσουν να μην εξυπηρετούνται στο μέλλον. Και δεν ξέρω αν αυτό μας συμφέρει. Όπως και να έχει, εάν δεν καλύπτεται στο πεδίο εφαρμογή αυτή τη πρόταση, πρέπει κάπως να τα αντιμετωπίσουμε. Και ε, υπάρχει το πρόβλημα, σιγά σιγά μειώνεται, αλλά όχι όσο γρήγορα θα έπρεπε. Τώρα, όσον αφορά την οδηγία, θα μπορώ να, μπορώ να είμαι πολύ σύντομη. Στην ουσία, η ανάκτηση των ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων και η ενίσχυση των ε, εγγυήσεων ε, θα πρέπει να δούμε αν θα γίνεται με εξοδικαστική διευθέτηση. Αυτό συμβαίνει σε περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, με βάση κάποιες δικλείδες ασφαλείας ή αν πρέπει να υπάρχει άλλη λύση. Θα ακούσω τις απόψεις σας από αυτού, θέλω να δω τι έχετε να πείτε. Αυτά λοιπόν, 7 λεπτά μήνυσα. Ρομπέρτο, νομίζω ότι αυτά ήταν τα βασικά θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν και προσβλέπω και ε, στις απόψεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ευχαριστούμε πολύ Έστερ. Και για την παρουσίαση. Πρώτα απ' όλα, φυσικά, να χαιρετήσουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες ε, συνάδουν και με το σχέδιο δράσης ε, του ΕΚΟΦΗΝ. Ακόμα και αν όλοι γνωρίζουμε ότι τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων σε πολλές χώρες είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει και επειδή τώρα ακριβώς έχουμε και την ε, ανάκτηση και επιπλέον ε, εποπτικές δυνατότητες, ε, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώνονται δραματικά. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι το να έχουμε ένα καλύτερο κανονιστικό πλαίσιο είναι η κατάλληλη κίνηση. Γι' αυτό και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε αυτές τις δύο προτάσεις και χαιρετίζω και το έργο που έχει κάνει μέχρι τώρα η Αυστριακή Προεδρία και ελπίζω να είστε σε θέση να ακολουθήσουμε παρόμοια προσέγγιση και για την ε, βελτίωση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι πολύ σημαντική για να καταφέρουμε να οριστικοποιήσουμε το φάκελο μέχρι το τέλος της θητείας να σταθώ μια στιγμή και ε, στον μηχανισμό προστασίας, στον backstop και με βάση τα όσα είπε και η Έστερ. Αντί να ξεκινήσουμε από συγκεκριμένε ε, επιλογές, θα ήθελα να αρχίσουμε με, με δύο βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το έργο μας. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει και για το Συμβούλιο. Η πρώτη αρχή Προφανώ υπάρχουν και διαφορέ και υπάρχουν στοιχεία συμπληρωματικότητας μεταξύ του πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Πρώτο πυλώνας έχουμε ένα υποχρεωτικό μηχανισμό προστασία, το backstop και το δεύτερο είναι ένα επιπρόσθετο ε, πλαίσιο που μπορεί να επιβάλλει η αρχή εποπτείας. που μπορεί να προσθεθεί ανατράπεζα. Όπως ξέρετε όλοι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή και το αντέντουμ της ΕΚΤ και ε, του Μηχανισμού Εποπτείας που είναι για τον πυλώνα 2 ε, σε ό,τι αφορά ε, τις προληπτικές προμήθειες βάσει των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο άρθρο 1 της CRD και η εξολόγηση των προμηθειών και πιθανή επιβολή επιπρόσθετων μέτρων αν θεωρηθεί ε, μη εύλογη η προσέγγιση από πλευρά υποπτία και οι δύο δραστηριότητε γίνονται ανατράπεζα, γιατί είναι μέτρο του πυλώνα 2. Πάνε λοιπόν στην τράπεζα, βλέπουν τι είδου έκθεση υπάρχει, λένε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν ε, επαρκούν οι λογαριασμοί και οι κανόνες ε, λογιστικών προτύπων. Πρέπει να κάνετε κάτι παραπάνω. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε από προληπτική άποψη. Αυτό είναι λογικό. Γιατί ξέρουμε ότι όλες, ε, όλα τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ε, πολλούνται με θετική αξία. Στην πράξη δηλαδή δεν συμβαίνει συχνά να είναι μηδενική η αξία. Μπορεί να είναι χαμηλή βέβαια η αξία, αλλά υπάρχει. Γι' αυτό και ο μηχανισμός αποπτείας λέει ότι θα φτάσει στο 100% μόνο αν για αυτά τα ανοίγματα υπάρχει μηδενική αξία. Γι' αυτό και είναι μέτρο του πυλώνα 2. Συμφωνώ με την Έστερ ότι μπορούμε να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, να ακολουθήσουμε την προσέγγιση των κατηγοριών ή μια διαφορετική προσέγγιση που θα εξηγήσω. Αλλά η πρώτη αρχή που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι ότι πρέπει να σεβαστούμε τη διαφορά μεταξύ υποχρεωτικού μηχανισμού πρόληψης backstop και πυλώνα 2 που ε, υιοθετείται και εφαρμόζεται κατά περίπτωση. Επομένω, πρώτα πρέπει να διαφυλάξουμε αυτή την διαφοροποίηση μεταξύ του πρώτου πυλώνα, που είναι υποχρεωτικό, δεσμευτικό, δεν εξετάζεται κατά περίπτωση, δεν αναλύουμε ούτε τι εγγυήσει ούτε τίποτα άλλο. Είναι τα βασικά που πρέπει να κάνει κάθε τράπεζα. Και επιπροσθέτω έρχεται ο δεύτερο πυλώνα, ε, που έχει τη διακριτική ευχαίρεια ο επόπτη να ε, επιβάλλει οι τράπεζες λοιπόν έχουν τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα εάν ε, η προσέγγιση που έχει ακολουθήσει η τράπεζα μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν επαρκεί. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαφοροποίηση. Αυτή είναι η πρώτη αρχή. Πρέπει να την τηρήσουμε. Αυτό γίνεται με διαφορετικούς τρόπου. Έχω προτείνει διάφορες ε, λύσεις. για να γίνεται σεβαστή αυτή η αρχή. Να διαβρύνουμε το χρονοδιάγραμμα. Ε, να έχουμε μεγαλύτερο χρονοδιάγραμμα για τα ε, μη ασφαλισμένα δάνεια. Όπου έχουμε μια περίοδο τριών, τεσσάρων, πέντε ετών. Νομίζω και τα κάτι μέλη τα συζητούν. Ή να έχουμε αντιθέτω το ίδιο χρονικό περιθώριο, αλλά υποχρεωτικά να έχουμε χαμηλότερο ποσοστό. Με τα 80, 90, 75% δεν έχει σημασία. Εγώ στέκομαι στην αρχή. Αυτό είναι η υποχρέωση που έχουν όλοι και μετά κατά περίπτωση ο, ε, ο SSM ή ο επόπτης που δεν είναι τραπεζική ένωση ε, συμπληρώνει το υπόλοιπο ποσοστό για να φτάσουμε στα 100%. Υπάρχουν ε, διάφοροι τρόποι λοιπόν από τεχνικής άποψης για να γίνει αυτό. Και για τα ασφαλισμένα και για τα μη ασφαλισμένα. Στην έκθεση FSC υπήρχε η ανεξάρτητη αξιολόγηση των εγγυήσεων. Τότε θεωρούμε ότι υπάρχει ε, η αξία. Άλλη επιλογή που εξετάζουν τα κράτη-μέλη να έχουμε ε, παράταση τη χρονική περίοδου. Άλλη επιλογή που ανέφερε η Έστερ είναι να μην είμαστε στο 100% αλλά με λίγο χαμηλότερο ποσοστό. Και μετά για τα μη ασφαλισμένα η υποπτική αρχή είναι που κατά περίπτωση αποφασίζει για να φτάσει στο 100%. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι από τεχνική άποψη να γίνει σεβαστή αυτή η αρχή και αυτό είναι απολύτω λογικό. Να υπάρχει διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Και βεβαίω και θέλουν να τα συζητήσουμε όλα αυτά από κοινού για να βρούμε τη σωστή λύση, που είναι κάτι πολύ δύσκολο. Έχουμε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα να έχουμε διάφορες κατηγορίες. Και μετά υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Είμαι διατεθειμένος να τα συζητήσουμε. Αυτό που δεν είμαι διατεθειμένος να συζητήσουμε είναι ότι ορισμού θα υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των δύο πυλώνων. Η δεύτερη αρχή τώρα. Βεβαίω και θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ δύο στοιχείων. Αφενό, να υπάρχει αυτή η σωστή ε, και αυτός ο εύλογος εφοδιασμός, ε, όμως ε, δεν θα πρέπει να υπάρχουν στρεβλώσεις και να αποφύγουμε τέτοια στρεβλά κριτήρια και κίνητρα για να οθήσουμε επιχειρήσεις προς την πτώχευση που θα μπορούσαν να σταθούν στην αγορά. Δεν θέλουμε λοιπόν να μορφώσουμε έναν μηχανισμό που ακριβώς επειδή είναι υποχρεωτικό για όλους, θα έχουμε την υποχρεωτική διάσταση. Και μετά όμως βλέπουμε ότι οθούμε προς τη χρεοκοπή επιχειρήσεις που μπορεί μόνο ένα τμήμα του ε, χρέους τους να ε, είναι αφαιρέγγιο. Αυτή είναι η δεύτερη αρχή λοιπόν που θα πρέπει να τηρήσουμε. Ένας τρόπος είναι αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ του going και του gone concern. Όταν λοιπόν ένας πιστολήπτης ε, δημιουργεί ε, πρόβλημα de facto ή ένας που ενδεχομένως δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν ε, θα πρέπει να τους οθήσουμε προς την χρεοκοπία όλους αυτούς. Και μετά έχουμε και την περίοδο χάριτος και το καθεξής. Ξέρω ότι και στα κράτη-μέλη υπάρχει αυτή η συζήτηση, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ε, τηρήσουμε αυτή την ε, αρχή. Για τα μη ασφαλισμένα, να προσθέσουμε μια περίοδο ενός ε, ή δύο ετών. Από τεχνική άποψη λοιπόν υπάρχουν πολλοί τρόποι, αλλά τουλάχιστον τώρα που βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια τη συζητηση πρέπει να συμφωνήσουμε επί τη αρχή περισσότερο να αποφύγουμε τα στρεβλά κίνητρα που θα εξωθούν ε, τις επιχειρήσεις και θα τις πρόχνουν εκτός αγοράς. Ενώ από την άλλη φυσικά θα πρέπει να έχουμε ε, τα απαραίτητα μέτρα που θα προστατεύουν ε, και τον τραπεζικό κλάδο υπό τον πυλώνα 1 και 2. Πήρα και τα δύο λεπτά που είχατε εξοικονομήσει εσείς. Σας ευχαριστώ. Και για την οδηγία βέβαια είναι πιο απλά τα πράγματα, αν και υπάρχουν ε, δυσκολίες. Ε, θέλουμε να ενισχύσουμε ε, το επίπεδο προστασίας από πιθανές καταχρήσεις. Όμως και πάλι το βασικό είναι ο κανονισμός. Εύχομαι και ελπίζω ότι αν παραμείνουμε σε επίπεδο αρχών υπάρχει περιθώριο συμβασμού. Όλοι λοιπόν σε αυτή τη βάση θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρεθεί κοινό τόπος. Είναι επίση σαφέ για μένα ότι αν δεν είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε έναν καλό κανονισμό, καλύτερα να μην έχουμε καθόλου. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Ευχαριστώ. Uh, okay. Now I wear back my head of chair. Επανέρχομαι στο ρόλο του Προέδρου. Σάντερ Λούνς, πρώτος κοιόδης. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Δύο λεπτά. Γιατί έχει και το ECR σκέδιο. Βεβαίω θέλω να γίνει αυτή η συζήτηση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, όπω απέδειξαν τα τελευταία αυτά λεπτά. Πρέπει να συζητήσουμε τα τεχνικά ζητήματα, τα μέσα. Και ο στόχος μας, ο στόχος πρέπει να επιτύχουμε είναι πολύ σημαντικός. Είπε και ο πρόεδρος ότι υπάρχει ζήτημα δημοτικότητα σε σχέση με τους ε, πολίτες. Αυτό πρέπει να επιτύχουμε. Και είναι πολύ πιο σημαντικό από τις συζητήσεις για τις ε, αρχές και τις ψήφους. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι κάποιες χώρες έχουν ε, δυσκολία να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ζητήματα και δυσκολίες στην ε, οικονομία τους, όπως είδαμε και με τα μια εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ιρλανδία. Υποστηρίζουμε τις ε, προσπάθειες ε, του SSM, συμφωνούμε με την Επιτροπή ως προς τον στόχο της αντιμετώπισης των υψηλών επιπέδων με εξυπηρετούμενων δανείων. Συμφωνούμε ταυτόχρονα ότι και εμείς ως νομοθέτες μπορούμε να συμβάλλουμε στη λύση. Η δεύτερη πρόταση του επεξηγηματικού υπομνήματος αναφέρει τη μείωση α, της ανάγκης να συμβάλλει στην ε, να συμβάλλει το κοινό, να επιβαρυνθεί το κοινό δηλαδή με τη μείωση των εξυπηρετούμενων ε, δανείων. Πρέπει λοιπόν να περιοριστεί η απώλεια κεφαλαίων από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτό το αναφέρει η κυρία Ντελάνγκε. Ταυτόχρονα όμως αυτή η έκθεση δεν αναφέρεται σε ισχύοντα σε τωρινά μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή έκθεση σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο μέλλον και σε αυτό πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Αυτό είναι ο προβληματισμό μου. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα καλύτερο για τη οικονομική σταθερότητα, δεν μπορούμε να στραφούμε προ το μέλλον περισσότερο. Ας κοιτάξουμε και αυτή την πτυχή λοιπόν. Με την τωρινή έκθεση με μια άλλη, δεν ξέρω αν ανοιχτό το ζήτημα, αλλά και η διαχείριση του κινδύνου έχει πολύ μεγάλη σημασία και για το υφιστάμενο ε, για τα υφιστάμενα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αντιλαμβάνομαι ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους αυξάνονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να ενισχύσουμε την ελάχιστη κάλυψη όπως πολύ σωστά λέει η έκθεση και παραθέτω αφού ύστερα από μερικά χρόνια δεν, καλύφθηκε, δεν χρησιμοποιήθηκε επαρκώς δεν θα πρέπει αυτή η κάλυψη να συνεχιστεί χωρίς να εξετάζονται τα αριθμητικά στοιχεία. Και για να ολοκληρώσω, γιατί είναι προκατακτικές μόνο οι παρατηρήσεις, θα ήθελα να κάνω και μια πολιτική τοποθέτηση. Γνωρίζουμε όλοι και αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα πολύ αμφιλεγόμενο κεφάλαιο και θα πρέπει πιστεύω να βρούμε κάποιες δημιουργικές συμβαστικές λύσεις. Ω και ο και εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στους ε, εισηγητές δηλαδή, είναι σημαντικό για μένα να ξέρω ότι δεν θα θέσουν σε κίνδυνο αυτή η συμβασμή τον ε, γενικό στόχο που είναι η μείωση του κινδύνου. Και γι' αυτό ιδιαίτερα θέλουμε να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου για την πτυχή αυτή. Πρέπει να γίνει σωστά αυτή η δουλειά, να λυθεί το ζήτημα πρώτα απ' όλα, πριν από τα υπόλοιπα θέματα και βεβαίως προσβλέπω στη συνεργασία με την συγκεκριτή και τους σκιώδεις. Και ευχαριστώ πολύ και για τον χρόνο που μου διαθέσατε. Ο κύριος Λούκε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα εστιαστώ στο δεύτερο, στη δεύτερη προσέγγιση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δηλαδή πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ε, διασφάλιση των πιστωτών και την αξιολόγηση. Η προσέγγιση της Επιτροπής με την νομοθετική της πρόταση νομίζω ότι μας επιτρέπει να προχωρήσουμε προς το στόχο μιας καλύτερα λειτουργούσας αγοράς για τις πιστώσεις με εναρμόνιση μέσω ελάχιστων προδιαγραφών και υπερσυνοριακή δραστηριότητα για τις επιχειρήσεις αυτές. Υποστηρίζω τους στόχους της πρότασης, ωστόσο θα ήθελα να διατυπώσω και τον εξής προβληματισμό ότι πρέπει κατά την αξιολόγηση της προσέγγισης να μιλήσουμε και το πεδίο των ε, μη εξυπηρετούμενων ε, δανείων. Είναι περιορισμένο αυτή τη στιγμή, δηλαδή πρόκειται για δάνεια τα οποία έχουν χορηγηθεί από ένα πιστοτικό ίδρυμα, έχουν αναλυφθεί από μη τραπεζικό ε, φορέα έτσι δηλαδή έχουμε να κάνουμε πιστώσεις ε, που δεν έχουν ε, εξαγοριστεί από τράπεζα ή δεν έχουν χορηγηθεί από μη πιστοτικό ίδρυμα. Εδώ λοιπόν πρέπει να έχουμε ένα level playing field, ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Και τα μέτρα τα οποία θα για ένα περιορισμένο αυτή τη στιγμή πεδίο, αλλά που θα πρέπει να ε, ανοίξουν σε ευρύτερο πεδίο της αγοράς, θα πρέπει να είναι μέτρα τα οποία δεν θα οδηγούν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Σε αυτό πρέπει να σταθούμε, πιστεύω ώστε να μην γίνει παρέμβαση τέτοια που θα, παρεμ... που θα ε, οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η υποτίμηση των ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων. Έτσι λοιπόν θα ήθελα με αυτές τις ε, πρώτες παρατηρήσεις, σε αυτές τις πρώτες παρατηρήσεις να σταθώ. Πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας μια συζήτηση που θα αφορά και τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις συνέπειες τους για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Κλείνοντας όμως θα ήθελα να κάνω την εξή ε, παρατήρηση για την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την εξουδικαστική ε, αξιολόγηση και τη βελτίωσή της, διότι εδώ είμαι επιφυλακτικός ως προς το εάν αρκεί η προσέγγιση αυτή, εάν μπορεί να καλύψει όλα τα προβλήματα. Τα εξοδικαστικά μέτρα για την ε, αξιολόγηση των εγγύσεων μπορεί να φέρουν αποτέλεσμα μόνο όταν υπάρχει αμφισβήτηση μεταξύ δανειολήπτη και δανειοδότη η Επιτροπή προτείνει να μπορεί να επανέλθει στα δικαστήρια αυτή η εξοδικαστική αξιολόγηση. Άρα ξανανοίγει το πεδίο της ε, ένδικης αμφισβήτησης. Μπορεί δηλαδή μια εξοδικαστική ε, λύση που αμφισβητείται να ξαναγυρίσει στα δικαστήρια για να διεκδικήσει τα δικαία του ενδιαφερόμενος. Ίσως ήταν όμως σωστότερο να παραιτηθούμε από την επιδίωξη μιας εξουδικαστικής αντιμετώπισης και να κοιτάξουμε να επιταχύνουμε τις δικαστικές διαδικασίες. Με αυτά κλείνω και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τους φιλελευθέρους ε, τώρα ο Ραμόν ε, Τρεμόσα Ιμπάτσελς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συζητητές, την Εστέρ Ντελάνγκε και τον Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη και τους συνεργάτες τους για τη δουλειά που κάνουν για αυτή την έκθεση και καλωσορίζω και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είμαι και ευχαριστημένος διότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ανάπτυξη που δείχνει ότι ε, μειώνεται το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα διάφορα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα στην Νότια Ευρώπη, ε, στην οποία υπήρχε ε, πριν από κάποια χρόνια ιδιαίτερο πρόβλημα με αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια. Έχουμε διαπιστώσει επίσης ότι αυτό έχει δημιουργήσει και ε, κάποιες ε, αντιπαραθέσεις, διότι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουμε κάποιες εκθέσεις οι οποίες λένε ότι λόγω του προβλήματος των κόκκινων δανείων σε κάποιες χώρες στην Νότια Ευρώπη δεν υπήρχε αρκετή δανειοδότηση από τις τράπεζες στην οικονομία και κάποιες ε, χώρες δεν αναπτύσσονταν όπως άλλες. Επίσης είδαμε και διάφορα έγγραφα από διάφορες κεντρικές τράπεζες σε εθνικό επίπεδο που λένε το αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ξέρω λοιπόν ότι το θέμα είναι ιδιαίτερος επίμαχο. Πριν αρχίσω λοιπόν να σας λέω τις απόψεις μου, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την ημέρα που ήρθε ο Μάριο Ντράγκ εδώ, σε μία ακρόαση στην ΕΚΟΝ τον περασμένο Νοέμβριο, και τον ρώτησα για την προέλευση αυτών των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και του είπα, κύριε Ντράγκη, εγώ είμαι της άποψης ότι είναι η έλλειψη εφαρμογής ε, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας Ιδέως ε, η οδηγία για τι καθυστερήσει των πληρωμών που είναι ε, στην πηγή των κόκκινων δανείων σε κάποιε χώρε. Και ο Μάριο Ντράκη είπε: Συμφωνώ πλήρω μαζί σα. Δεν είναι μόνο οι πολυεθνικέ οι οποίε δεν πληρώνουν τι μικρομεσαίε ε, επιχειρήσει που το 2008-2009 προκάλεσαν αυτή τη μαζική ανεργία γιατί δεν πλήρωναν. Και κάποιες κυβερνήσεις επίσης για χρόνια δεν κατέβαλαν τα δεδουλευμένα σε, μικρο, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε μέτρα για να αποφύγουμε μελλοντικέ κρίσει με εξυπηρετούμενο ε, δανείων. Γιατί σε κάποιε χώρε δεν υπάρχει κυφεστό κυρώσεων εάν μια πολυεθνική δεν πληρώνει τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα μου και θα επανέλθουμε σε αυτό. Επίσης, είμαστε της άποψης ότι πρέπει να υπάρχουν και κάποιες ε, διατάξεις ε, όταν τα δάνεια αρχίζουν να μην εξυπηρετούνται. Βλέπουμε πόσο διαφορετικά αντιδρούν τα κράτη-μέλη, πόσο διαφορετική νομοθεσία χρειάζεται μια κάποια εναρμόνιση. Αλλά επίση πρέπει να λάβουμε υπόψη και ότι έχουμε τελείω διαφορετικά τραπεζικά συστήματα. Για παράδειγμα, στην Νότια Ευρώπη, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία έχουμε ε, συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα και 4-5 μεγάλες τράπεζε έχουν το 80% τη αγορά, ενώ αντιθέτω, βλέπουμε στη Βόρεια Ευρώπη Υπάρχει ένα μοντέλο, το οποίο κατά την άποψή μου είναι καλύτερο. Υπάρχουν κάποιες μεγάλες τράπεζες, οι οποίες δραστηριοποιούνται και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και εκατοντάδες μικρές ε, τράπεζες αποταμιευτικές. Και άκουσα διάφορες απόψεις από διάφορους αδέλφους, από διάφορες ομάδες, από διάφορες χώρες που λένε ότι χάρη σε αυτό το δίκτυο των μικρών αποταμιευτικών τραπεζών Όταν υπήρξε η κρίση των subprime, ε, κατάφεραν να σώσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έτσι δεν είχαμε μαζική ανεργία. Σώσαμε τις επιχειρήσεις, σώσαμε θέσεις εργασίας, σώσαμε τις κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι και αυτή μια άποψη και πρέπει να τα λάβουμε και αυτά υπόψη, ότι υπάρχουν διαφορετικά τραπεζικά συστήματα στην Ευρώπη και γι' αυτό και αντιλαμβάνομαι και την άποψη του Προέδρου Γκουαλτιέρη που είπε ότι δεν μπορούμε να έχουμε αρκετά καλή νομοθεσία, είναι καλύτερο να μην έχουμε νομοθεσία. Εγώ ελπίζω ε, ότι θα βρούμε αυτή την καλή νομοθεσία γιατί είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα σε κάποια κράτη-μέλη. Καλό τις δύο μεγάλες ομάδες να καταλήξουν σε συνένεση και οι φιλελεύθεροι είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν και να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια νομοθεσία η οποία θα επιτρέψει σε επόμενη κρίση μια εξυπηρετούμενο δανέο να μην είναι τα πράγματα τόσο δραματικά όσο στο παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Ραμόν. Ο Σβεν Γίγκολτ. Ναι. Ο Ερνέστο Τασούν και εγώ είμαστε συνεισηγητές, συν σκιώδεις θα μιλήσω λοιπόν πρώτα για τον κανονισμό. Είναι σαφές ότι τρόπον την η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί μια σταδιακή προσέγγιση και αυτό δείχνει και μια κάποια σοφροσύνη, αλλά δεν αγγίζει τους πιο ευαίσθητους τομείς. Τα παλιά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, και εγώ από δημοκρατική σκοπιά το βρίσκω μάλλον δύσκολο για να το θέσω έτσι. Γιατί σημαίνει ότι η αντιμετώπιση των παλιών κόκκινων δανείων de facto αφήνεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Ευρωζώνη, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει νομοθεσία από αυτόν και τελικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφασίζει πώς θα ρυθμιστούν. Ε, αυτό δεν άρεσε στην ομάδα μου, είναι γνωστό Α, πώς ε, εσείς, ε, ακόμα και εσείς κύριε Πρόεδρε που σας εκτιμούμε ιδιαιτέρως, ασχοληθήκατε με το θέμα αυτό. Τώρα λοιπόν είναι η ευκαιρία ο δημοκρατικός χώρος να νομοθετήσει επ' αυτού. Και θα υπάρχουν προβλήματα αν δεν τα καταφέρουμε. Υπάρχει βέβαια και μια μέση οδός, να πούμε ότι όσον αφορά τους ορισμούς, θα μπορέσουμε να πάμε πιο κοντά στα όσα προβλέπει η ΕΚΤ που περιλαμβάνει περισσότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παρά το γεγονός ότι δεν αγγίζει καν τα παλιά δάνεια και τα αφήνει σε μία εξέταση ένα περίπτωση του πυλώνα 2. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βεβαίω φοβήθηκε ε, να έχει μια πάρα πολύ σαφή πολιτική για το θέμα γιατί είναι λεπτό. Αλλά τουλάχιστον θα μπορούσαμε να διευρύνουμε πολύ πιο εύκολα το πεδίο εφαρμογή έτσι. Και πέραν αυτών περιμένω να δω και τι θα προκύψει με τη συζήτηση μεταξύ μας. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ακολούθησε τη συμβουλή τη ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συνοδεύεται και μία, μία εντολή δηλαδή αυτή η υποχρεωτική προληπτική στάση για να δούνε ποια δάνεια θα μπορούσαν να καταλήξουν να είναι μη εξυπηρετούμενα. Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε να, ε, να δεχτούμε. Επίσης υπάρχουν επιπλέον πιέσεις να μειωθεί το επίπεδο των κόκκινων δανείων είτε μέσω νομοθεσίας είτε μέσω ε, της έκτη μέσω δράσης εποπτείας. Να μπορέσουμε να πιέσουμε δηλαδή τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια στον κόσμο των σχεδόν τραπεζών και των ανοιχτών χρηματοπιστωτικών αγορών που πιέζουν προς ε, μεγάλες εκπτώσεις ε, σε σχέση ε, με την σωστή τιμολόγηση αυτών των δανείων. Μέχρι τώρα 18 από τα 28 κράτη-μέλη ε, εξετάζουν, έχουν τη δυνατότητα να, να συσταθεί μια κακή τράπεζα. Θυμάμαι και την πρόεδρο τη CBA που είπε ότι αν δημιουργηθεί πλαίσιο για κακές τράπεζες θα ήταν ε, ένα τρόπος να ζητούμε ευρωπαϊκές λύσεις. Ξέρω ότι ο πρόεδρος ποτέ δεν μπόρεσε να εξηγήσει επακριβώς πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε απλώς τη μετατόπιση της ευθύνη ε, προς το έναν ευρωπαϊκό χώρο. Αλλά εν γέννη έχει δίκιο. Ε, χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο για τις κακές τράπεζες. Και τέλος θα ήθελα να τονίσω και λυπούμαστε ότι διότι η ρηστικοποίηση της Βασιλείας 3 χρησιμοποιεί την προσέγγιση της εσωτερικής αξιολόγησης που επιτρέπει να έχουμε 0% επιτόκιο σε τέτοια στοιχεία αποθεματικού ε, και γιατί δεν το έχει κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν το έχει ρυθμίσει. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με λίγα λόγια για την οδηγία. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι καλή ιδέα να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός κανονισμός και να υπάρχει ένα πλαίσιο για να έχουμε μια καλύτερη ευρωπαϊκή αγορά, η οποία θα έχει τραπεζική ένωση. Αλλά στην πρόταση δεν υπάρχουν εύρωστοι κανόνες για την προστασία των καταναλωτών και το ελάχιστο επίπεδο το οποίο επιλέγεται κατά την άποψή μας δεν αντανακλά επαρκώς το γεγονός ότι αν δοθεί ένα δάνειο σε ένα καταναλωτή ουσιαστικά ξεκινάει και μια κοινωνική σχέση αμοιβαία υποχρέωσης. Εάν το πουλήσει, ακόμα και αν διαφωνείτε κύριε Λόκε, εγώ πιστεύω τις χριστιανικές κοινωνικές ε, ηθικές αξίες. Δηλαδή, μια κοινωνική σύμβαση δεν είναι απλώ μια χρηματοπιστωτική σύμβαση, είναι απλώ μια, και μια συμφωνία μεταξύ διαφόρων παραγόντων. Που σημαίνει ότι εσύ δεν πρέπει να ξεπουλά τον πελάτη σου ε, διότι ο πελάτη συνειδητοποιεί ότι αύριο μπορεί να μην είναι πελάτη τη τοπική του τράπεζα στην Ισπανία, αλλά πελάτη ενό hedge fund που εδρεύει κάπου αλλού, σε τελείω διαφορετικό μέρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό το θέμα και ακόμα και αν ε, καλωσορίζουμε την πιο ευρωπαϊκή και καλύτερη λειτουργία της αγοράς, θα πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και οι καταναλωτές θα πρέπει να κάνουν μια συνειδητή επιλογή. Θέλουν στο μέλλον να μπορεί να πληρωθεί το δάνειό τους ή θέλουν να αποκλείσουν αυτό το ενδεχόμενο. Και αυτό δεν θα πρέπει ε, να βρίσκεται στα ψηλά γράμματα μια σύμβαση. Θα πρέπει να είναι μια συνειδητή επιλογή και μπορεί κάποιο να πρέπει να πληρώσει και κάποιο αντίτιμο αν δεν θέλει να ξεπουληθεί το δάνειό του. Αυτή θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παπαδημούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, συζητούμε ένα πολύ σημαντικό φάκελο και με την πρόταση για τον κανονισμό και με την πρόταση για την οδηγία. Πρώτα απ' όλα από το μέγεθος του προβλήματος. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγγίζουν το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ και επηρεάζουν και την πορεία της οικονομίας των κρατών μελών και επομένως της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλούν την υγεία του τραπεζικού συστήματος σε ένα ενδεχόμενο μιας νέας κρίσης και συνδέονται και με την παγωμένη συζήτηση για το περίφημο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων, τον περίφημο τρίτο πυλώνα, για τον οποίο δεν έχουμε κανένα νέο ουσιαστικό και καμία πρόοδο ουσιαστική. Και σε αυτό έχει ευθύνη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί ο σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της Ευρωμάδας Αριστεράς για το θέμα του έντις έχω να ακούσω νέα από την Εστέρ Ντελάγκε που είναι η εισηγήτρια εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Πιστεύω λοιπόν ότι ως Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να προσπαθήσουμε με τις αναγκαίες συζητήσεις, με τους αναγκαίους συμβιβασμούς και μεταξύ μας να οθήσουμε σε μια προσπάθεια να υπάρξει μια ευρωπαϊκή εναρμόνιση, να υπάρξουν κάποιοι κανόνες, να ενισχυθούν, παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, ε, δεν μπορώ έτσι, it's impossible to speak. να υπάρξουν κάποιοι κανόνες που να προστατεύουν τους καταναλωτές και να δούμε πώς θα δημιουργηθεί ένας υποχρεωτικός μηχανισμός προστασίας, αυτό το περίφημο backstop, και πώς θα υπάρξει και ένας δεύτερος συμπληρωματικός πυλώνας, τον οποίο θα τον χειρίζονται μέσα σε ένα πλαίσιο σαφό, ε, σαφές κανόνων, ο αρμόδιος φορέας για την εποπτεία, ο SSM. Νομίζω ότι αν αποτύχουμε και αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν και πάμε και αφήσουμε και αυτούς τους φακέλους για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, μετά τις προσεχείς ευρωεκλογές, θα είναι πάρα πολύ αρνητικό. Πιστεύω ότι είναι λάθος η θεωρία πρώτα θα μηδενίσουμε τον κίνδυνο και μετά θα αρχίσουμε να συζητούμε για τον επιμερισμό του. Αυτά τα πράγματα πρέπει να πάνε παράλληλα και όσο πιο αποτελεσματικοί είμαστε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο να γίνουν κάποια βήματα με αφορμή αυτούς τους δύο φακέλους για τη μείωση των κινδύνων θα βοηθήσουμε και στο να προχωρήσει το ίντις αλλά και να προετοιμαστεί το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα από την κρίση που θα έλθει. Γιατί οι κρίσεις κάνουν κύκλους. Και αν θέλουμε να μπορούν οι τράπεζες να δίνουν δάνεια για να τροφοδοτούν επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για να δίνουν στεγαστικά δάνεια σε νέα νοικοκυριά που θέλουν να αποκτήσουν ένα σπίτι, για να βοηθούν startups, πρέπει να βρούμε κανόνες που να βοηθήσουν με έναν ε, τρόπο συμφωνημένο οπωσδήποτε να μειωθούν αυτός ο όγκος, ο, ο, μεγάλος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και εδώ επιτρέψτε μου να έχω μια διαφορετική γνώμη από τον κύριο Λούκε. Πιστεύω ότι και η μέθοδος του εξοδικαστικού συμβιβασμού και της αναζήτησης εξοδικαστικών λύσεων στο να βρίσκονται λύσεις σε αυτά τα θέματα βοηθά γιατί πολλές φορές μόνο η αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης πολλές φορές δημιουργεί υπερβολικές καθυστερήσεις και ε, γραφειοκρατία ε, και δεν βοηθά ε, στο θέμα αυτό. Επειδή από τη συζήτηση προκύπτει Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Προκύπτει πολύ μεγάλο έδαφος για συζήτηση, συνεννόηση και αναζήτηση συμβασμών στη συνεργασία μεταξύ των σκιωδών εισηγητών. Περιμένουμε ενδιαφέρον από τους δύο συνεισηγητές συγκεκριμένες προτάσεις ή δυνατόν και που να συμφωνούν μεταξύ τους έτσι ώστε και εμείς να μπορέσουμε με τις τροπολογίες να συμβάλλουμε στη συζήτηση αυτή που είναι πάρα πολύ σημαντική. Um, e uh, ευχαριστώ, Μάρκο Βαλή, η e FTD. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όπως και ο Δημήτρης Παπαδημούλης, θέλω και εγώ να εστιάσω τη συζήτηση στο θέμα του επιμερισμού του κινδύνου, δεδομένου ότι η εισηγήτρια και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πολύ σωστά επισημαίνει την ανάγκη να περιοριστεί ο κίνδυνος. Ωστόσο ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό και να προχωρήσουμε παράλληλα έτσι ώστε να υπάρξει περιορισμός και αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στο θέμα αυτό. Βεβαίως έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα ως προς τον ε, κίνδυνο για τις τράπεζες των ε, ρευστών και παράγωγων τίτλων. Και εδώ έχουμε μια πρώτη αξιολόγηση του SSM που αναμένεται. Πρέπει να είμαστε θέση λοιπόν αυτή οι ρευστή τίτλοι που ανέρχονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κυρίως για τα χαρτοφυλάκια, για κάποιες, κάποιων ιδιαίτερα σημαντικών για το σύστημα τραπεζών. Πρέπει λοιπόν να βρούμε και για αυτούς κάποιες λύσεις αποτελεσματικές που μπορεί να φαίνονται απόμακρες αυτή τη στιγμή για περιόδους που θα είναι ίσως ε, λιγότερο ταραγμένες. Γιατί βλέπουμε ότι μπορεί να χάσουν σε περιόδους κρίσεως ε, σημαντικό μερίδιο της αξίας τους αυτή η Πρέπει και σε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει λύσεις ώστε να εξασφαλιστεί διαφάνεια στο θέμα αυτό. Για την δέσμη των μη εξυπηρετούμενων ε, δανείων συμπερίζομαι τις προτάσεις του συναδέλφου Δημήτρη Παπαδημούλη, επίσης τα όσα είπαν οι πράσινοι για την εποπτεία και προστασία των, καταναλ... Ε, ε, πολιτών που έχουν των καταθετών αλλά και την ανάγκη προστασίας γενικότερα της οικονομίας όπως υπόθηκε ήδη. Πιστεύω ότι πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα στο ζήτημα των ε, ε, κερδοσκοπικών ταμείων, ώστε να μην κινδυνεύσει και η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και πρέπει να δοθούν λύσεις που να προστατεύουν τον καταθέτη, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα επιβίωσης του ίδιου του οικονομικού συστήματος μέσα στην Ευρωζώνη. Ας μην είμαστε λοιπόν υπερβολικά επιθετικοί με μια πολύ βιαστική και γρήγορη λύση η οποία θα μπορούσε και να μην αντιμετωπίσει τα ζητήματα της κερδοσκοπίας αλλά και να θέσει κερδίρο τον καταθέτη και όποιον, έχει, όποιον διακρατά τέτοια ε, στεγαστικά δάνεια. Ώστε να μην περάσουν αυτά μόνο σε εκείνους που θέλουν να κερδοσκοπήσουν. Πρέπει να έχει βεβαίως τη δυνατότητα και την υποχρέωση ο δανειολήπτης να αποπληρώσει το δανειό του μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα κατά προτίμηση εναντί εκείνου ο οποίος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αγορά βλέπουμε ότι αναπτύσσεται μια ε, παράγωγη αγορά ταχύτατα και βεβαίως πρέπει να ε, τοποθετηθούν η Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διάφοροι οργανισμοί με ε, δημόσιες τοποθετήσεις. Πρέπει τις επόμενες εβδομάδες να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Υπάρχουν σημεία σύγκληση είμαι βέβαιος, σε πολλά θέματα και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λύση που θα προβάλλει το Κοινοβούλιο για να μην περιοριστούμε μόνο σε κάποιες ενδείξεις που δεν είναι και σωστές απαραίτητα. Ευχαριστώ. Τσάνι. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους δύο συντάκτες για τις ε, παρεμβάσεις τους. Είναι σαφές ότι δεδομένη τη σημασία ε, του θέματος, τα θέματα τα οποία είπατε είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά, υπάρχουν διαφορετικά οράματα και θέσει, ανάγκες και επιλογές αναλόγω των διαφόρων κρατών μελών. Σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και γενικά το τραπεζικό σύστημα στην ε, Ευρώπη, σε σχέση με το ενεργητικό αυτό έχει γίνει πολλή λόγο. Ίσως να μην έχουμε αρκετά εστιαστεί στα πραγματικά νούμερα και βέβαια στις συνέπειες τους και στις βαθύτερες αιτίε που μας έφεραν στην κατάσταση αυτή. Ίσως δεν χρειάζεται τόσο αφηρημένη ανάλυση. Ανάλυση που θα μιλά για συνθήκες αγοράς, για τραπεζικά συστήματα με συμπεριφορά ή διαχείριση αδιαφανή. Γιατί πάνω απ' όλα το ξέρουμε, το έχουμε δει όλοι, τα αίτια της κατάστασης τα τελευταία 8-9 χρόνια που αντιμετωπίσαμε τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση της Υπήρου μας ε, στην σύγχρονη ιστορία της, μας φέρουν ενώπιον ε, στοιχείων αριθμητικών και δεδομένων που φέρνουν σε πολύ δύσκολη κατάσταση στις τράπεζες σε σχέση με μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Γίνεται λόγος και εδώ λοιπόν για την μείωση του κινδύνου, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και τα νούμερα. Είδαμε την έκθεση σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια πολλών τραπεζών, όλο και πιο υψηλή εκθετικά ε, αυξανόμενη έκθεση που περιορίζεται τα τελευταία δύο χρόνια καθώς ε, έχει αρχίσει σιγά σιγά η ανάκαμψη. Πολλές τράπεζες και μάλιστα πάνω απ' όλα μεγάλα πιστοτικά ιδρύματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν αγορε, ε, τιμές αγοράς ή τιμές που ορίζουν οι μεγάλοι ε, παράγοντες που δραστηριοποιούνται στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ε, πρέπει λοιπόν τώρα να κοιτάξουμε ποιος πραγματικά δεν είναι σε θέση να ανθέξει τόσο χαμηλές τιμές και αναγκάζεται να διατηρήσει την έκθεση. Σε αυτό θα πρέπει να εστιαστούμε. Αυτή είναι η ουσία της συζήτησης στα δύο αυτά θέματα αλλά πάνω απ' όλα με τις ρυθμίσεις αυτές δεν πρέπει να πέσουμε στον κίνδυνο να δημιουργήσουμε ένα νέο μεταγενέστερο πρόβλημα ή να εκθέσουμε σε νέες δυσκολίες ένα ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα το οποίο ήδη αντιμετωπίζει πολύ σημαντικά προβλήματα. Πολύ σημαντικό για τα θέματα αυτά θα είναι να επαληθεύσουμε ότι, να βεβαιωθούμε ότι αφενός μεν η όποια ρύθμιση για την πώληση πακέτων μη, κυβερνη... μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και η κάλυψη, το πλαίσιο κάλυψης των απολειών να μην φέρουν αρνητικές συνέπειες, δεσμενείς συνέπειες για τους ε, διάφορους παραγόντες και τις τράπεζες. Ενδιαφέρον επίσης θα είναι να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο για τις ε, asset management corp companies, επιχειρήση διαχείριση ενεργητικού, για όποιον δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει την εξέλιξη των τιμών ε, και δεν μπορεί ω εκ τούτου να πωλήσει ή να ρευστοποιήσει ε, πακέτα με εξυπηρετούμενων δανείων. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχει κάποια κάλυψη μέσω ενός ρόλου που θα πρέπει να αναπτύξουν και τα ίδια τα κράτη-μέλη. Ένα μοντέλο για αυτές τις επιχειρήσεις διαχείρισης ενεργητικού με συνεργασία μεταξύ κρατικών αρχών και τραπεζών και ιδιωτικών ε, φορέων. Αυτή θα είναι η πραγματική πρόκληση. Και το τελευταίο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ, που ήδη όμως τόνισαν αρκετοί συνάδελφοι, έχει να κάνει με την ε, ταχεία διαδικασία για τις εγγύησεις. δεδομένου ότι δεν είναι ισότιμοι οι όροι ε, κυρίως ενημέρωσης, πληροφόρησης που έχουν οι διαφοροί παράγοντες, δανειολήπτες, δινοδότες, τραπεζικά ιδρύματα κτλ. Πάνω απ' όλα πρέπει να σταθούμε στην προστασία του καταναλωτή. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ε, έχω άλλα αιτήματα στη διαδικασία του Κάτστη. Uh, Η Εστέρ παρακαλώ. Um, uh, τέσσερα λεπτά ο καθένας. Ευχαριστώ, δεν θα χρειαστώ εγώ τέσσερα λεπτά. Η συζήτηση πήγε προς την κατεύθυνση που περίμενα να πάει. Δεν χρειάζεται λοιπόν να πούμε και πολλά, θα τα συζητήσουμε όλα. Θα ήθελα να πω ε, κάτι για την, αυτή τη συζήτηση όλη για την πίεση προς την αφαιρεγγιότητα. Δεν θα ήθελα να συγχαίουμε ένα αίτημα για αρκετές δικλείδες ασφαλείας ως μια πίεση προς ε, ερεγγιότητα. Έχουμε διάφορα μαξιλαράκια, έτσι παίζεται το παιχνίδι και τα χρειαζόμαστε γιατί το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο. Τώρα το θέμα της εξοδικαστικής ρύθμισης. Δεν είχαμε τόσο πολύ χρόνο να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Είναι αμφιλεγόμενο μεν, αλλά πρέπει να πω κύριε Λούκε ότι αν δεν συζητήσουμε το θέμα της εξοδικαστικής ρύθμισης, όπως είπατε, και προσπαθήσουμε απλώς να επιταχύνουμε τις νομικές διαδικασίες, προς το παρόν δεν ε, έχουμε καταφέρει να προχωρήσουμε την όλη συζήτηση για την περιορισμένη εναρμόνιση της νομοθεσίας περί Αφού δεν προχωρούν λοιπόν όλα αυτά, δεν θα ήθελα τώρα να χάσουμε και τη δυνατότητα της εξοδικαστικής ρύθμισης, που λειτουργεί αποτελεσματικά σε αρκετές χώρες μέλη. Πολύ ευχαρίστω να το συζητήσουμε, αλλά η εναλλακτική σας πρόταση δεν νομίζω να μας ε, ε, οδηγεί και πουθενά γρήγορα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της εξοδικαστικής ρύθμισης και την προστασία των καταναλωτών, Συμφωνώ για την ανάγκη να υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, αλλά σας παρακαλώ συνάδελφοι διαβάστε τι έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα καταναλωτικά δάνεια και τα ενυπόθηκα εξαιρούνται από ε, αυτή την πρόταση. Διορθώστε με αν πιστεύετε αν υπάρχει ένα παραθυράκι αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι τα περισσότερα καταναλωτικά προϊόντα, τα στεγαστικά δάνεια είναι τα πιο σημαντικά, εξαιρούνται από την πρόταση. Να τα δούμε λοιπόν, να τα συζητήσουμε. Λειτουργεί σε αρκετά κρατημέλη. Α μην χάσουμε λοιπόν και αυτή τη δυνατότητα. Ευχαριστώ συνάδελφοι για τη συμβολή σα. Πάρα πολύ χρήσιμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Εστέρ. Και εγώ θα ήθελα να είμαι σύντομο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω απλώς σε κάποια σχόλια. Η πρώτη προς τον κύριο Σάντερ. Δεν νομίζω ότι το να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε ανεπιθύμητες συνέπειες ε, ε, είναι πρόβλημα δημαγωγίας, είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Επομένως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι το οποίο Ε, να μην μας οδηγήσει σαν επιθύμητες συνέπειες και να το ανακαλύψουμε κατόπιν εορτής. Θέλουμε κάτι το οποίο να είναι αξιόπιστο και ε, να λειτουργεί προληπτικά. Νομίζω ότι ο Σβέν Γκίγκολτ έκανε μια σημαντική παρατήρηση όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή ε, του θέματος. Αλλά νομίζω ότι όταν θέσατε την ερώτηση, ουσιαστικά απαντήσατε μόνο σας. Εάν θέλετε να αντιμετωπίσετε από νομοθετική σκοπιά στο όλο θέμα του αποθεματικού, δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα απλώς με ένα χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να κάνουμε αυτό που πρότεινες, δηλαδή να έχουμε τη φιλοδοξία να συζητήσουμε τα στοιχεία, να δούμε πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συστημική λύση για το πρόβλημα με τις κακές τράπεζες, με τις ευρωπαϊκές αρχές κλπ. Εγώ είμαι ανοιχτό ε, καταρχήν. Πιστεύω, λαμβάνοντας υπόψη και τη χρονική συγκυρία και τις διάφορες ε, θέσεις ε, στο Συμβούλιο και μεταξύ των μελών εδώ στο Κοινοβούλιο. Δεν θα το καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε, αλλά θα το μετανιώσουμε και συμφωνώ μαζί σας εδώ ότι το καλύτερο θα ήταν να επιδείξουμε το απαραίτητο σθένος, να προτείνουμε κάτι πιο ε, συνολικό. Και εγώ ε, επικροτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνολική προσέγγιση, αλλά ξέρουμε όλοι ότι η οδηγία από μόνη της δεν αρκεί για να δημιουργήσει μια αγορά. Και το σχεδιάγραμμα ούτως ή άλλως μας δείχνει ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ ήπιο νομοθέτημα, το οποίο απλώς περιγράφει την παρούσα κατάσταση. Πρόκειται λοιπόν για μια άγουσα που για διάφορους λόγους δεν ε, επελέγει και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι θα πρέπει να σεβαστούμε και το πεδίο εφαρμογή ε, το οποίο καθορίστηκε και το σχέδιο δράσης ε, του ΕΚΟΦΗΝ και προτάθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι εξήγησα σαφώς τις δύο αρχές. Και πάλι, Έστερ, σίγουρα δεν θα πρέπει να ε, ε, πιέσουμε τις, τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να υπάρχει κίνδυνος προς αφαιρεγγιότητα, αλλά δεν θα πρέπει επίσης να παριστάνουμε και ότι δεν υπάρχει. τα κράτη-μέλη συζητούν διάφορες λύσεις για να λάβουν υπόψη και τις περιπτώσεις τις οποίες ε, έχουμε μία πλήρη ε, έκθεση. Πώς θα την ορίσουμε, πώς θα κάνουμε τη διάκριση ε, μεταξύ της going concern και της gone concern. Εγώ είμαι ανοιχτό στη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται στο σχέδιο πρότασης είναι πολύ περιορισμένος. Και ελοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε έκθεση που λαμβάνεται υπόψη σε περιπτώσεις που είναι μόνο τμήμα της έκθεσης μια μικρομεσαίας επιχείρησης που κατά τα άλλα είναι βιώσιμη και το υπόλοιπο κομμάτι μπορεί να παραμείνει στην αγορά. Ε, ουσιαστικά γίνεται όλο το δάνειο μη εξυπηρετούμενο και τελικά πολλέται και σε κάποιον, επομένω δεν υπάρχει καμία ευκαιρία ανάκτηση των κονδυλίων και τελικά διώχνουμε από την αγορά ένα σημαντικό σκέλος της οικονομίας μας. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι, ότι ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος και πρέπει να δούμε με ρεαλιστικό τρόπο πώς μπορούμε να δώσουμε την πιο σωστή απάντηση. πρέπει ταυτόχρονα να είμαστε και δίκαιοι, αλλά να το κάνουμε και με απλό τρόπο. Εγώ λοιπόν είμαι ανοιχτός σε συμβιβασμούς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, αλλά όπως σας είπα, εξακολουθώ να θεωρώ ότι τα δύο βασικά θέματα που ανέφερα, δηλαδή ότι ο πυλώνας 1 ε, δεν μπορεί να είναι το ίδιο με τον πυλώνα 2 και ότι αυτές οι πιθανές ανεπιθύμητες ε, παρενέργειες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, είναι τα βασικά κεντρικά στοιχεία της συζήτησής μας. Ε, είδα ότι όλη η διαπραγματευτική ομάδα ασχολείται με το θέμα αυτό. Θα μπορούσε λοιπόν να είναι ένα σημείο εκκίνωσης, παρά τη διαφωνία, και νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα μπορούμε να συζητήσουμε και ή δυνατόν να καταλήξουμε και σε μια συμβαστική και βιώσιμη λύση. Αλλιώς, όπως σας είπα, αυτή είναι και η άποψή μου, δεν υπάρχει ε, κανονισμός που να είναι καλύτερος από κακό κανονισμό. Καλό είναι να μην έχουμε τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Θα βρούμε μια καλή λύση. και θα προχωρήσουμε λοιπόν την νομοθετική μας εργασία σε θέματα μείωσης κινδύνου. Χρονοδιάγραμμα τώρα. 22 Οκτωβρίου εξέταση σχεδίου έκθεσης, προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών 26 Οκτωβρίου. Όντως είναι λίγο σφιχτό το χρονοδιάγραμμα, θα το συζητήσουμε. Εξέταση των τροπολογιών 19 και 20 Νοεμβρίου, ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ 3 Δεκεμβρίου. Νομίζω ότι πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα πέραν ε, το θέμα των τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ την Έστερ και όλους εσάς ε, για αυτή την ε, πολύ πλούσια και χρήσιμη πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα που όπως γνωρίζετε δεν είναι οι ψηφοφορίες αλλά μια πολύ σημαντική εκλογή. Εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου διότι όπως θα ακούσατε, στις 29 Αυγούστου η ομάδα του ΕΛΚ εξέλεξε τον Μάρκους Φέρμπερ ως ε, τον νέο συντονιστή της ΕΚΟΝ. Καταρχάς λοιπόν να συγχαρούμε τον Μάρκους Φέρμπερ και μετά από την επιλογή του αυτή ο Μάρκος παρετήθηκε από πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΕΚΟΝ, επομένως τώρα θα εκλέξουμε τον νέο πρώτο αντιπρόεδρο. Καταρχάς πρέπει να σας πω ποιοι αναπληρωτές συμμετέχουν στις πληροφορίες βάσει των κανόνων μας. Η Σαμπίνε Βερχάιεν, ο Κρίστοφ Χάνσεν, ο Ραμέν Χουαρέγγι, ο Μπράντο Μπενιφέη, Άσλι Φόξ, Σόφι Ίνεντβελτ, Παλώμα Λόπες Μπερμέχο. Καταρχάς να επαληθεύσουμε την απαρτία. 16 μέλη, ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να σας ζητήσω να ορίσουμε τους υποψηφίους για πρώτο αντιπρόεδρο. Ο Λούντεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος του ΕΛΚ θα ήθελα να προτείνω τον κύριο Μπράιαν Χέις. Ευχαριστώ. Δέχεται ο υποψήφιος την υποψηφιότητα. Ναι κύριε Πρόεδρε, τη δέχομαι. Ωραία και ξέρω ότι ο υποψήφιος είναι πλήρες μέλος της Επιτροπής ΕΚΟΝ, ξέρω ότι ε, έχει κάνει και τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων, επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκλογή διαβοής. Συγχαρητήρια. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Λούντεκ και τους συναδέλφους που με έθεσαν υποψήφια για αυτή την πολύ σημαντική θέση. Όποιες και αν είναι οι πεπιθήσεις μου ε, για διάφορα ζητήματα και οι απόψεις μου για διάφορα ζητήματα που συζητήθηκαμε, συμφωνούμε ότι για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας, μέσω της συνεργασίας ε, θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε με όλους τους αντιπροέδρους ε, και ιδίως με εσάς κύριε Πρόεδρε, προβλέπω σε αγαστή συνεργασία με όλους σας. Ευχαριστούμε, Μπράιον. Και εμείς ε, περιμένουμε να αρχίσουμε τη συνεργασία μας. Ωραία. Θεωρούμε ότι έχει εκλεγεί ο υποψήφιο διαβοή. Παρακαλώ, ελάτε εδώ. Α, α, κατάλαβα. Καλύτερα να μείνετε εκεί, κατ' εξαίρεση αυτή τη φορά. Ο πρώτος ε, αντιπρόεδρος δεν θα καθίσει εδώ στο Προεδρείο, αλλά και πάλι συγχαρητήρια, Brian. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Πρώτα, ας ελέγξουμε έναρξη ψηφοφορίας. couple of colleagues to vote. Want to vote yet? Please. Is it test. Vote. Who is not voting? Who has put the voting card? Ψηφίζουμε δοκιμαστικά, παρακαλώ, λείπουν ορισμένοι συνάδελφοι. Εντάξει, δεν είναι και υποχρεωτικό. Πέρας. Just a second. So we close the vote. Thank you. So now, uh, we uh, start... Ωραία. Θα περάσουμε στην πολύ σημαντική ψηφοφορία του επόμενου ζητήματο. Πρόταση κανονισμού. Ναι, το είδα. Για το πανευρωπαϊκό ατομικό δεξιοδοτικό προϊόν, η συγγήτρια η Σοφία Νιτφέλτ, η Περβάνς Μπερές θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία για αυτή την πρόταση που είναι πολύ σημαντική ε, στην νομοθετική δέσμη που έθεσε επιτάπητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατανοώ ότι όλοι θέλουν να ε, ξεκινήσουν και πάλι διαδικασίε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο, το Συμβούλιο Δυνατών, για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Πρόκειται για μια σημαντική πρόταση με στόχο τη δημιουργία ενός ε, νέου ε, στεξιωτικού συστήματος για το σύνολο των Ευρωπαϊκών πολιτών. Δεν υπήρξε συζήτηση στην ε, Επιτροπή για αυτό που θα ψηφίσουμε. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Φαντάζομαι ότι και η συγγήτρια θα θέλει να τοποθετηθεί από πλευρά τη. Θα μπορούσε και να ψηφιστεί τον Ιούνιο το κείμενο βέβαια, ίσως να ψηφιστεί σήμερα. Για τη δική μας πολιτική ομάδα, έχουμε ε, και τα διάφορα, τις διάφορες ιδιαιτερότητες ε, των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κάθε πολιτική ομάδα τελικά πήρε τη θέση της, αλλά εμείς ε, μόλις σήμερα το απόγευμα μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια θέση για το τελικό κείμενο πριν από την συνεδρίαση σήμερα. Εντάξει, δεν θέλω να σταθώ στα επιμέρους ηχεία προβληματισμού των ΜΕΝ και των ΔΕ, αλλά θα ήθελα να θίξω τα εξή. Πρώτον, για το ζήτημα της αρμόδιας αρχής που διαχειρίζεται αυτά τα προσωπικά προϊόντα. Ε, εδώ υπάρχουν ορισμένες αρμοδιότητες που εκχωρούνται στην ΕΣΜΑ. Υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες σε ό,τι αφορά την ελεύθερη ε, παροχή υπηρεσιών, σε ό,τι αφορά τις συντάξεις. Μετά έχει να κάνει και με το πολιτικό μήνυμα ότι μία η σωστή αρμόδια αρχή είναι ο ΑΙΟΠΑ και όχι η ΕΣΜΑ σε ό,τι αφορά τι συντάξει. Αυτό όμω ε, βλέπουμε ότι υπάρχει στην πρόταση των συμβαστικών προτάσεων. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τον ορισμό του κεφαλαίου. Υπάρχει ο κίνδυνο, ο ορισμό που προτείνεται εδώ στο 2.21 άρθρο, να μην επιτρέπει στου συνταξιούχου να έχουν πρόσβαση στο σύνολο ε, του κεφαλαίου που έχουν αποταμιεύσει. Και αυτό είναι σφάλμα. Γι' αυτό και θέλαμε, τελευταία στιγμή το ξέρω, αλλά πρέπει να υπάρχει και κάποια κατανόηση, ένα περιθώριο ευελιξίας, ειδικά σε ένα τόσο ευαίσθητο φάκελο. Κάναμε λοιπόν μια ε, προφορική ε, τροπολογία που θα την υπενθυμίσουμε και στη συνέχεια, αλλά την παραθέτω τώρα θέλαμε να πούμε ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για μία ε, προφορική τροπολογία των πρασίμων για την οποία θα θέλαμε να ε, πάρουμε το λόγο συγκεκριμένα. Ευχαριστούμε πολύ. Σοφή, θες να πάρεις το λόγο? Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδεις και το επιτελείο που έχει εργαστεί πολύ σκληρά το τελευταίο χρόνο. Ο φάκελος αυτός ε, και το τελικό κείμενο είναι πολύπλοκο αλλά ιδιαίτερα ισορροπημένο και τελικά είναι μια συμβαστική πρόταση. Ξέρω ότι είναι λεπτό το ζήτημα, αλλά αυτό που πετύχαμε εδώ πραγματικά ε, αξίζει τη στήριξη όλων και όλων των πολιτικών ομάδων. Γιατί όλες οι πολιτικές ομάδες ε, κατάφεραν να αποσπάσουν ε, πολλά μέσω των τροπολογιών τους. Οι διαπραγματεύσεις για τις ε, τροπολογίες πήραν πολύ καιρό. Αρχικά είχαμε σκοπό να, τα, ψηφίσουμε την πρόταση τον Ιούνιο. Ε, ανεβάλλει η ψηφοφορία ακριβώς για να έχουμε δύο παραπάνω μήνες, να τα συζητήσουμε και στις πολιτικές ομάδες. Ξανακαθίσαμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. καταλήξαμε στη συμφωνία την περασμένη Τρίτη. Οι συμβιβαστικές προτάσεις ε, κυκλοφόρησαν την Τετάρτη το πρωί και συμφωνώ βέβαια με την Περβάνς Μπερές ότι πάντα πρέπει να υπάρχει ευελιξία στη διαδικασία και να λαμβάνουμε υπόψη και προτάσεις της τελευταίας στιγμής. Από την άλλη όμως ε, υπάρχει και το ζήτημα της διαφάνειας στη διαδικασία. Το να δίνουμε δηλαδή τη δυνατότητα στους συναδέλφους ε, και το χρόνο να απαντήσουν και να εξετάσουν νέες ιδέες και προτάσεις. Οπότε τώρα ένα νέο στοιχείο, το οποίο δεν έχει θυγεί καθόλου τον τελευταίο χρόνο. Ξαφνικά σήμερα το απόγευμα ε, μπαίνει ε, στην όλη συζήτηση ως προφορική τροπολογία. Εντάξει, δεν ξέρω, το σημειώνω, ας ψηφίσουμε. Ελπίζω οι σοσιαλιστέ και δημοκράτε να είναι σε θέση να στηρίξουν την πρόταση όσο έχει για να αρχίσουμε τι διαπραγματεύσει στη συνέχεια του μήνα και να ολοκληρώσουμε, ελπίζω, μέχρι τα τέλη τη χρονιά. Και πάλι, ω εκπρόσωπο ε, κεντρώου κινήματο, θεωρώ ότι πρέπει να πούμε και να γνωρίσουμε ότι είναι μια ε, πολύ ισορροπημένη συμβαστική πρόταση, καλύπτει όλε τι πολιτικέ ομάδε, είναι πιο ευρωπαϊκή, δίνει καλύτερη προστασία του καταναλωτή, καλύτερες ευκαιρίες ε, για του παρόχου. πολλά στοιχεία βιωσιμότητας, ε, κοινωνικής ευθύνης και ούτω καθεξής. Πραγματικά είναι μια σφαιρική πρόταση που αξίζει τη στήριξή σας. Ελπίζω όσο γίνεται περισσότεροι συνάδελφοι να τη στηρίξουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Brian. Ναι, ένα σύντομο σχόλιο εξ ονόματος του ΕΛΚ, Πρόεδρε. Θέλω να συμφωνήσω με την εισηγήτρια για αυτό το ζήτημα. Ήταν δύσκολη η διαπραγμάτευση, ε, περίπλοκη και όλες οι πολιτικές ομάδες έχουν επιδείξει ευελιξία για να καταλήξουμε ε, σε αυτή την καταλητική πρόταση την τελευταία εβδομάδα και η ομάδα μου με εξοδότησε να στηρίξω αυτή την πρόταση βάσει αυτών που σας προανέφεραν και βάσει του κειμένου που διανεμήθη την περασμένη εβδομάδα. Είναι πολύ αργά πλέον να εισάγεται μια τροπολογία τώρα ε, που ούτε προτάθηκε ποτέ και ούτε συζητήθηκε ουσιαστικά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό και υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που επιτρέπει και προβλέπει ένα συγκεκριμένο όριο υποβολή τέτοιων τροπολογιών. Πέραν τούτου, όλε οι πολιτικέ ομάδε έχουν συμβιβαστεί για να καταλήξουμε σε αυτή την πρόταση και για τη δική μα πολιτική ομάδα υπάρχουν στοιχεία που δεν μα ικανοποιούν. Όμω, εφόσον πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό προϊόν και όπω είπατε και εσεί, Πρόεδρε, είναι ε, αναπόσπαστο τμήμα της, του θεματολογίου τη Ένωση των Κεφαλαγορών, ε, είναι βασικό στοιχείο για το μέλλον των Ευρωπαίων πολιτών. Έχουν γίνει λοιπόν και από τον ΑΕΟΠΑ συγκεκριμένα σημαντικές ε, υποχωρήσεις. Ε, η ΑΕΟΠΑ είναι βασική αρχή που ασχολείται με την συνταξιδοτική πολιτική. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία μου δημιουργούν πρόβλημα, αλλά τα δέχτηκα στο πνεύμα συμβασμού. Και για τον ορισμό του κεφαλαίου. Νομίζω ότι τώρα έχουμε έναν ορισμό που ευσταθεί στην πράξη, ε, μπορεί να λειτουργήσει και μπορεί να έχει ε, καλά αποτελέσματα και για τους ε, πολίτες αλλά και για τον ανταγωνισμό, με διαφάνεια πάντα. Όλοι υποχώρησαν λοιπόν, όλοι συμβιβάστηκαν. Αλλά το ξαναβάζουμε ένα στοιχείο τόσο τελευταία στιγμή. Όταν οι συνάδελφοί μου μου έχουν δώσει την εξουσιοδότηση και μου έχουν δώσει το πράσινο φως να το υπερψηφίσω, είναι πρόβλημα. Και ήθελα να το επισημάνω πριν την ψηφοφορία. Ευχαριστούμε πολύ. πώς θα λύσουμε αυτό το ζήτημα μόνο για της ψηφοφορίας. Μόνο έτσι θα λυθεί δημοκρατικά. Για τις ε, τρεις τροπολογίες λοιπόν ε, θα ξεκινήσουμε με από κοινού ψηφοφορία για τις τροπολογίες 177, 178 και 179 που ζητούν την απόσυρση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ουσιαστικά και αν υιοθετηθούν δεν θα υπάρξει περαιτέρω ψηφοφορία. Βέβαια, αν απορριφθούν οι τροπολογίες, δεν θα καταγραφεί το αποτέλεσμα ε, της ψηφορίας στην τελική έκθεση. Ήταν κάτι που έπρεπε να διαβάσω. Ωραία. Ψηφοφορία από κοινού τροπολογίες 197 έως 199. Υπέρ. Ηλεκτρονικά. Α, με ονομαστική κλίση. Έναρξη. Vote is Πέρας. Απορρίπτονται. Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική β με προφορική τροπολογία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ο κ. Λούκε. Συγγνώμη, αλλά αντιτίθεμε σε αυτή την τροπολογία. Ρωτήστε αν αντιτίθεται κάποιος άλλος, γιατί δεν την έχουμε δει καν αυτή την τροπολογία. Ωραία, να τη διαβάσω, την τροπολογία, για λόγους διαφάνειας. Να προσθέσουμε το κεφάλαιο σημαίνει αθρηστική συνεισφορά και επιστροφή σε αυτές τις, ε, συνεισφορές, στις υπόψη το σύνολο το, του κόστους ε, και τον τελών και ούτω καθεξής. σημαίνει ότι υπάρχει επιστροφή μόνο όταν έχουμε θετικέ τιμέ και όχι αρνητικέ. Και δεύτερον, παραπέμπει στον ορισμό στο άρθρο 37 για να εξηγήσω. Έχετε ένσταση. Τέσσερι ενστάσεις χρειάζομαι. Εντάξει, υπάρχουν. Απορρίπτεται λοιπόν η προφορική τροπολογία. Να ψηφίσουμε επί της συμβιβαστικής. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Όχι, δεν ετίθεται στη ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, ψηφίζουμε για τη συμβαστική Β με ονομαστική κλίση. Γίνεται αυτό, εφόσον ε, το ζητούν οι σοσιαλιστές. Επομένω, ψηφίζουμε για τη συμβαστική Β με ονομαστική κλίση. Έναρξη. Πέρας. εγκρίνεται 22 υπέρ, 4 κατά, 21 αποχές. Συμβαστική γάμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική δέλτα, υπέρ, κατά, α, συγγνώμη και εδώ υπάρχει η προφορική τροπολογία των πρασίνων. Δεν υπάρχουν ενστάσει. Μαζί με την προφορική λοιπόν. Α, υπάρχει ένσταση. Ο κύριος Λούκε. Ναι, ένσταση γιατί δεν γνωρίζουμε ποια είναι η τροπολογία. Α, δεν τη γνωρίζετε. Διαγραφή του σημείου F του άρθρου 5 παράγραφος 1 Δεν την έχω εγώ στον κατάλογο ψηφοφοριών. Εντάξει, εντάξει. Μπας. Ε, δεν ξέρω τι κατάλογο ψηφοφοριών έχει ο συνάδελφο. Υπάρχει σε όλου του κατάλογου ψηφοφοριών. Έχει αποσταλεί από την περασμένη εβδομάδα και στου Κιώδη. Είναι κάτι τελείω διαφορετικό από την προφορική τροπολογία των σοσιαλιστών. Επομένω, ε, δεν ξέρω πώς ε, δεν υπάρχει στον κατάλογο ψηφοφοριών του ECR και, στη δική μου, και στο δικό μου κατάλογο υπάρχει, λέει ο πρόεδρο, και στον κατάλογο του Elk. Μπέρντ, τη βρήκε. Εντάξει. Ε, φυσικά, αν έχετε αντίρρηση μπορείτε να το λέτε, αλλά όχι λέγοντας ότι είναι κάτι που δεν γνωρίζετε. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει. Φυσικά και μπορείτε να υποβάλλετε ένσταση αν θέλετε. Λοιπόν, υπάρχει ένσταση. Όχι. Συμβαστική δέλτα λοιπόν μαζί με την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε χωρί την προφορική τροπολογία, λοιπόν, τη συμβαστική δέλτα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε. Μπορούμε να ελέγξουμε, παρακαλώ, για τη συμβαστική δέλτα. Ε, ήταν σαφές το αποτέλεσμα, αλλά εντάξει. Άρχεται η, συμβασ... η ψηφοφορία για τη συμβαστική δέλτα. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε ψηφίσαμε. Τώρα πάμε στην ε, α. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σίγμα Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 535 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Συμβαστική 536. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 90. Υπέρ, κατά, ας ελέγξουμε την 90. Πέρας. Απορρίπτεται. 95 της ΙΜΚΟ. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 95 της ΙΜΚΟ. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 26 υπέρ, 23 κατά. Συμβαστική M. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. N. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική π με προφορική τροπολογία που δεν είναι καινούρια. Υπέρ κατά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Έγκρινεται. 24 υπέρ, 22 κατά. Τρεις εποχές. Συμβαστική Q. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική R. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική S. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική TAF. Υπέρ, α, Συμβαστική TAF με προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά. Ας ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψηφοδιαφορά. Ψηφίζουμε λοιπόν για τη σημαστική ΤΑΦ χωρίς την προφορική. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. V υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. X υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ΑΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ΑΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία Α αποσύρεται. Οπότε, σημαστική ΑΔ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σημαστική ΑΕΦ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 138 της ΣΥΜΚΟ, υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. 670 υπέρ, κατά, νομίζω απορρίπτεται, ας ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφορία για την 670. Πέρας. Απορρίπτεται. AG, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. AH, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AI και AK υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. AJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σημαστική 704 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε για την 704. Vote is closed. Πέρας. Απερίφθη. Με δύο ψήφους διαφορά. 25-23. AL συμβαστική υπερκατάποχες εγκρίνεται. Συμβαστική AM υπερκατάποχες εγκρίνεται. 631 και 903-905 αμπλοκ μπλοκ κατά επαληθεύουμε Πέρας. απεριευθεί ΑΕΛ συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 1 έως 8 υπέρ κατά επαληθεύμα. Ένα, δύο, οχτώ, εκατόν είκοσι οχτώ. Έμπλ δεν χρειάζεται να επαληθεύσουμε. Πέρα τη ψηφοφορία απερίφθη 158 ΙΜΚΟ υπέρ. Καλά, επαληθεύουμε. 158 ΙΜΚΟ. Πέρας. Και εγκρίνεται. 26 υπέρ 23 κατά συμβαστική AO υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΕΙΠ συμβαστική με προφορική τροπολογία των πρασίνων υπέρ κατά αποχές απερίφθη επαληθεύουμε αρχίζει η ψηφοφορία πέρας 19 υπέρ 30 κατά συμβαστική 80 χωρίς την ε, προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική AQ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται AR υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική AS υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ASA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται AT συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται AU συμβαστική υπερκαταποχές εγκρίνεται AV συμβαστική υπερκαταποχές εγκρίνεται AW συμβαστική υπερκαταποχές εγκρίνεται AX συμβαστική υπερκαταποχές εγκρίνεται AY υπερκαταποχές συμβαστική υπερκαταποχές εγκρίνεται AZ συμβαστική υπερκαταποχές εγκρίνεται BA συμβαστική υπερκατά εγκρίνεται BB συμβαστικη υπερκατα κατά επαληθεύουμε πέρας εγκρίνεται Α94 όχι 93 όχι, δεν έχει αποσυρθεί. Ε, A93 υπέρ κατά. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά αν θέλετε επαληθεύουμε. A93. Πέρας. Απερίφθη. A93, 94, ε, όχι ταυτόσημη, 95, υπέρ κατά αποχές συμβαστική BC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 298 με 292 υπέρ κατά επαληθεύουμε παρακαλώ πέρας απερίφθησαν Συμβαστική BD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 167 68 τη ΣΥΜΚΟ υπέρ. Καλά, ας επαληθεύσουμε νομίζω ότι εγκρίθηκαν. Πέρας. Εγκρίθηκαν. 26-22 ε, συμβαστική BE υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 913 υπέρ κατά επαληθεύουμε 913 πέρας απεριφθεί 914 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επαληθεύουμε 9-14 αρχίζει ψηφοφορία. 9-1-4. 9-14. Έχω θετικό πρόσημο στον καταλογό μου εγώ. Γι' αυτό και θεώρησα ότι εγκρίνεται. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 180 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Έμπλ 1 υπέρ εγκρινεται Πέρα τη ψηφοφοριας εγκρινεται 180 υπερ κατα αποχες απεριφθη εμπλ 1 υπερ κατα επαληθεύουμε. Πέρας. Απερίφθη. BF συμβαστική υπερκατά αποχές εγκρίνεται. 180 υπερκατά αποχές απερίφθη. ΜΚΟ 2 υπερκατά εγκρίνεται. 186 στην επόμενη σελίδα 186 το βρήκατε υπέρ κατά αποχές απερίφθη 187 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 191 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 192 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 3 υπέρ όχι επαληθεύουμε πέρας και εγκρίνεται 25 υπέρ 23 κατά 193 τώρα υπέρ κατά αποχές απερίφθη 196 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 194 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 199 υπέρ κατά αποχές απερίφθη έμπλη 5 υπέρ κατά επαληθεύουμε Πέρας. Απερίφθη έμπλ 7 υπέρ κατά. Αποχές απερίφθη. 8 έμπλ υπέρ κατά. Αποχές απερίφθη. 9 της έμπλ υπέρ κατά. Αποχές απερίφθη. 10 της έμπλ υπέρ κατά. Αποχές απερίφθη. 11 της έμπλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 της έμπλη υπέρ κατά αποχές επερίφθη 2002-08 απερίφθη 209 ε, ε, υπέρ κατά αποχές απερίφθη 5 υπέρ κατά αποχές και επαληθεύουμε πέρας και απερίφθη 6 της ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές απερίφθη εγκρίνεται συγγνώμη 7 της ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 της ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές απερίφθη BG συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 212 υπέρ κατά αποχές και δεν βλέπω να σηκώνω τα χέρια. Επαληθεύουμε 212. Πέρας. Απερίφθη 213 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 214 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 217 υπέρ κατά Επαληθεύουμε. 217. Και έμπλου 14. Πέρασε. Απερίφθη. 218 υπερκατάποχες. Απερίφθη. ΥΜΚΟ 6 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. ΥΜΚΟ 9 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 10 ΥΜΚΟ εγκρίνεται, 11 τη Ήμκο απερίφθη. 219 υπέρ κατά επαληθεύμα, 219. Πέρας εγκρίνεται 26 υπέρ 23 κατά και πάμε στη 222 και 14 τη ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 τη ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές απερίφθη 13 τη ΣΥΜΚΟ υπέρ και ελέγχουμε πέρας απερίφθη 17 της ΕΜΠΛ υπέρ κατά αποχές απερίφθη 16 της ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε αρχής προφορία πέρας 23 υπέρ 22 κατά εγκρίνεται 223 και 7 υπέρ κατά επαληθεύουμε Απερίφημε απερίφθη μία ψήφο διαφορά 25-24 ΙΜΚΟ 15 υπέρ και επαληθεύουμε Πέρας. Εγκρίνεται. 26 υπέρ, 23 κατά. 8 υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθη 226 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη 227 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη 17 της ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 228 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 9 υπέρ κατά επαληθεύουμε πέρας απερίφθη 229 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 230 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 231 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 18 της ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές απερίφθη 23 της ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά ας επαληθεύσουμε πέρας απερίφθη 26 υπέρ 23 κατά 19 της ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές απερίφθη 232 19 έμπλ είπε τα σχόλια δεν ακούγονται 232 και 19 αυτό είπα έχετε κάποια αντίρρηση ψηφίσαμε την ΕΜΚΟ 19 και έμπλη 19 232 έμπλη 19 αυτό είπα υπέρ Κατά επαληθεύουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 233 συμβατή υπέρ. Κατά. Αποχές περίφθη 234 έμπληκωση 20 υπέρ επαληθεύουμε πέρας Απερίφθη 235 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 236 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 237 υπέρ κατά επαληθεύουμε τη 237 πέρας απερίφθη 238 υπέρ κατά επαληθεύουμε τη 238 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απερίφθη. 20 της ΣΥΜΚΟ υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. Πέρας. Απερίφθη. 12 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 239 υπέρ κατά επαληθεύουμε πέρας απερίφθη 240 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 21 τη ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές απερίφθη 241 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 242 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επαληθεύουμε 242 άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 28 2.42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.44 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 245 υπέρ. Κατά επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 2.45. Πέραση της ψηφοφορίας. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τα μέλη της ΛΥΜΠΕ δεν μπορούν να ψηφίσουν, εκτός και αν είναι πληρωτές ε, της ΕΚΟΒ. Εκεί βεβαίως μέχρι να φτάσουμε στο συγκεκριμένο αριθμό. Μπορούν να ψηφίσουν με αρκεί να μην αλλάζει η ισορροπία της ομάδας. Έχουμε μέλη ε, της ΛΥΜΠΕ που δεν είναι αναπληρωτές. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν με τον αριθμό. Δεν ξεκίνησε ακόμα η κοινή συνεδρίαση. Μπορούμε να ψηφίσουμε μέχρι το όριο φυσικά. 2.46 Υπέρ Κατά Αποχές Απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 22 της έμπλη υπέρ κατά αποχές δεν βλέπω τίποτα. Ψηφίζουμε την 22 της έμπλη. Άρχεται η ψηφοφορία. Ακόμα δεν έχουν ψηφίσει όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά συμβαστική τροπολογία BH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, απορρίπτεται. 2.55 και έμπλη 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.56 υπέρ κατά επαλήθευση της 256 άρχεται η ψηφοφορία. We are reaching the limit. Now we are 61, but still. Colleagues can vote. Now... Έχουμε έναν επιπλέον τώρα. Γιατί δεν δείχνει τις ομάδες. Έχουμε μία επιπλέον ψήφο. No, no, but, but uh, actually there are the actual votes, so they are the register, so that's why it works. Sorry, it can work because actual vote is 50. Λειτουργεί το σύστημα. Μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε τις ψήφους πέρα τη ψηφοφορίας. Εντάξει, είναι λίγο ασυνήθιστο. Έχουμε ισοπαλή, επομένως απορρίπτεται. Ήμκο 27 τώρα, υπέρ. Κατά. Επαλήθευση της ΥΜΚΟ 27, άρχεται η ψηφοφορία. Ελπίζω να μας δείξει τις ομάδες. Τώρα έχουμε τρεις επιπλέον από τους σοσιαλιστές. Τρεις. Ένας επιπλέον. Εντάξει τώρα, πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 2.57 και έμπλη 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 258 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 259 υπέρ Εγκρίνεται, επομένω πάμε στην 261 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλη 28 υπέρ, κατά, επαλήθευση της έμπλο 28, αμπλοκ με τη 262 και τη 263 και την 29 της έμπλων. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 264 υπέρ. Υπέρ το ΕΛΚ. 264 υπέρ. Κατά επαλήθευση της 264 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση έρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ήμκο 30. Όχι εγκρίνεται, άρα καταπίφτει οι υπόλοιπε 266 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 31 ΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 32 υπέρ κατά επαλήθευση της ΕΜΠΛ 32 άρχεται ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. 27 όλα απορρίπτεται. Ήμκο 32 που είναι συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλη 23 υπέρ κατά θα την επαληθεύσουμε αυτή, M23, κατά πάσα πιθανότητα απορρίπτεται, αλλά να δούμε. Πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 25-30. Η συμβαστική BHA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2,70 και ΙΜΚΟ 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 36 υπέρ κατά αποχές δεν βλέπω εδώ σε αυτή την πλευρά να το επαληθεύσουμε λοιπόν έρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται έμπλη 33 υπέρ κατά επαλήθευση της ΕΜΠΛ 33, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οι υπόλοιπες καταπίπτουν. Η 2.72 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική BI υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 278 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 279 υπέρ κατά επαλήθευση της 279, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 281 υπέρ κατά Μάλλον έχουμε την ίδια ψηφοφορία. Επαλήθευση για την 281 παρόλα αυτά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία. 280 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 έμπλο και 282 υπέρ. Κατά Επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική BJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική BK υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 και 2,92 υπέρ κατά. Α, ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Περνάμε στη 294. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω αρκετά χέρια. 294. Ελέγχουμε. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται, συμβαστική BL υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ΙΜΚΟ 41 υπέρ κατά επαλήθευση της ΙΜΚΟ 41, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 303. Um, 303 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Πέρας ψηφοφορίας. Ισοπαλία. Απορρίπτεται. 304 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 42 ΙΜΚΟ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική BLA υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, έμπλη 43 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 23 υπέρ, κατά, επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας, απορρίπτεται, έμπλη 44 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική BM υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική BN υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 47 υπέρ κατά επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ήμκο 48 υπέρ. Το ΙΣΙΑ είναι κατά σε αυτή την περίπτωση. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική BO υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά επαλήθευση 24 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 312 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 312. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ήμπο 49 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλη 48 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3.19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 και 49 της έμπλου υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3.20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3.21 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική BQ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 και ΙΜΚΟ 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν ξέρω αν θέλετε να επαληθεύσουμε. Επαλήθευση. Πέρας ψηφορίας εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Καλά κάναμε και ελέγξαμε. 31 ΙΜΚΟ 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 323 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 324 και έμπλη 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 326 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 327 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, έμπλου 51 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 328 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, έμπλου 52 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, έμπλου 53 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, έμπλου 54 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 50 υπέρ κατά αποχές. Ήμκο 54 έχετε δίκιο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι υπόλοιπε καταπίπτουν, επομένως πάμε στην έμπλη 55. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3.30 καταπίπτει, Επομένω ψηφίζουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίας εγκρίνεται 29 ψήφοι υπέρ, 10 κατά, 17 αποχές. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 176 στο νομοθετικό ψήφισμα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε για την απόφαση να ξεκινήσουν οι διοργανικές διαπραγματεύσεις με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία και για τη σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία 47 υπέρ, 8 κατά και μία εποχή. Έχουμε την απαραίτητη ειδική πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Yes. So, uh... Uh, Έχουμε καθυστερήσει λίγο. Θα αλλάξουμε λοιπόν τη σειρά. Πάμε κατευθείαν στην ψηφορία Econ για να μην σας κρατήσουμε εδώ. Και μετά θα μας μείνουν μερικές ακόμα μόνο για για την εικόνα. Γιατί κάθεστε τόσο μακριά μου.